Dear colleagues, please take your seat. Καθίστε. Herzlichen Dank. Σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που σήμερα έχουμε μεταξύ μας ε, τον ε, εκπρόσωπο της ΚΝΕΣΕΤ, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, με τους συναδέλφους του από διάφορες ε, ομάδες. Είχαμε ήδη ενδιαφέρουσες συζητήσεις και νομίζω ότι είναι μια χρονική στιγμή επικαιρή και ότι είναι κάτι το οποίο ταιριάζει με τις συζητήσεις μας σήμερα το πρωί με τους ανθρωπικού Εξωτερικών του Ιράν. Και διαπιστώνουμε ότι το θέμα της Μέσης Ανατολής μας ενδιαφέρει όλους και ότι υπάρχουν αλλαγές στην περιοχή οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις και στο Ισραήλ. Μεταβήκαμε και μια, με μια αποστολή στην Αίγυπτο και είδαμε ποιες είναι οι συνέπειες και από την άλλη πλευρά αυτό ισχύει και για το Ισραήλ και παράλληλα ανησυχούμε για κάποιες συζητήσεις οι οποίες διεξαγάγονται και όπου μας δίνεται η αίσθηση ότι η λύση των δύο κρατών η προϋπόθεση της οποίας αποτελεί ε, βάση για τις μελλοντικές συζητήσεις δεν έχει τόσο πολλές πιθανότητες ε, ενδεχομένως και θα πρέπει λοιπόν να επαναφέρουμε και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και την το κύρος ε, των ελευθερικών διαπραγματεύσεων, ε, γιατί και αυτό θα αποτελούσε σταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή. προκειμένου να διευκολυνθεί και η διαδικασία. Σήμερα λοιπόν το πρωί συνομιλήσαμε με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών και η σχετική συμφωνία την οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική γιατί θεωρούμε ότι η πυρηνική εξέλιξη του Ιράν α, καθίσταται πιο δύσκολη, αυτό είναι φαντικό. και ασκήσαμε και κριτική στο ρόλο του Ιράν του πολέμου για αντιπροσώπου στη Μέση Ανατολή. Και δείξαμε και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Δεν είμαστε λοιπόν ε, μονοπλευροί, ούτε τυφλοί, δεν εθελοτυφλούμε. Και θα θέλαμε να συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την καλή συνομιλία, γιατί πέρα από την κριτική την οποία ασκούμε και για την Ισραηλινή πολιτική, όπως άλλωστε και οι Ισραηλινοί ασκούν, πολιτική, ασκούν κριτική στην πολιτική μας, κοιτώντα το υπόλοιπο συγκείμενο, αν θέλετε, της περιοχής, το Ισραήλ είναι η μοναδική δημοκρατία. Έτσι είναι. Δεν ξέρω στην ε, γειτονική περιοχή να υπάρχουν άλλες δημοκρατίες. Και πέρα λοιπόν από την κριτική που ασκούμε υπάρχει επί της αρχής μια συμπάθεια προς το Ισραήλ. Ο κύριος Χάνεκ λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είστε επί πολλά έτη φίλος της ε, χώρας και πολλές φορές φιλικά μας ε, επικρίνετε και μας ε, εξηγείτε τις απόψεις σας με κάποιο τρόπο αρκετά αποφασιστικό, ευθύ αλλά και φιλικό. Οπότε γι' αυτό και εμείς δεχθήκαμε αυτή σας την πρόσκληση να έρθουμε σε αυτήν την τόσο σημαντική συνάντηση και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε μια μοναδική ευκαιρία σε διάλογο, ούτω ώστε να δούμε κάποια ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά για την Ευρώπη αλλά και για το Ισραήλ και να δούμε και ε, διάφορα τα οποία ε, μας κένα για να βρούμε κάποιες απαντήσεις. Οπότε έχουμε μια αντιπροσωπεία από τον συνασπισμό που έρχεται στην ε, αντιπολίτευση. Α, εδώ είναι ο κύριος ε, Μιχαήλ, το εργατικό κόμμα που είναι ο κομματικός προϊστάμενος του δοσιπίν της ε, αντιπολίτευσης Μαστίγιο σημαίνει WIP, δεν το κρατάει το μαστίγιο, αλλά δίνει μάχες πραγματικές κατά της ε, κυβέρνηση. Σήμερα όμως ήρθε μαζί μας αυτή την σημαντική επίσκεψη. Ο κύριος Γιάκοφ Πέρι, επίσης, άλλος φίλος, που επί πολλά έτη υπηρέτησε στις υπηρεσίες ε, ασφαλείας, ε, επίσης ε, υπουργός τεχνολογίας και επιστήμης. Τώρα και αυτό συμμετέχει στην Προεδρία, ο κύριος Γιακόμπ, ο οποίος ήταν ο πρέσβης μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει συγγράψει μια σειρά βιβλίων και είναι πάρα πολύ σημαντικό μέλος της Επιτροπής μας και επίσης ε, συμμετέχει και αυτός στον συνασπισμό ε, που ονομάζεται Κούλαν, συνασπισμό κομμάτων. Οπότε εμεί τώρα εδώ αισθανόμαστε ότι είμαστε εν μέσω της οικογένειας μας ε, γιατί και εμείς συμμεριζόμαστε τις αξίες τις ευρωπαϊκές, συμμεριζόμαστε τις ελπίδες σας, τις φιλοδοξίες σας και αυτό αφορά το ιδεολογικό επίπεδο. Γιατί ξέρετε οι, οι γονείς προέρχονται από την Ευρώπη, οι γονείς και οι παππούδες, για άλλους από την Πολωνία, για άλλους από την Ελβετία, για άλλους από την Ουκρανία και την Πολωνία. Ο δικός μου πατέρας γεννήθηκε στην Πολωνία. Οπότε έχουμε μία σειρά Ισραηλινών ή μάλλον τους περισσότερους των Ισραηλινών που θέλουν να αναβαθμίσουν τις ε, σχέσεις της χώρας μας με την Ευρώπη. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε τι θα πει selfie. Selfie είναι όταν κανείς παίρνει φωτογραφία του εαυτού του, το selfie. Αλλά selfie σημαίνει και κάτι άλλο. Είναι η περιοχή που ζούμε, Συρία, Αίγυπτος, ε, ε Λίβανος, ε, χώρα των Φιλιστέων και Ιράν. Σέλφι, τα, τα αρχικά είναι οι χώρες που μας περιβάλλουν οι χώρες, οπότε πολλές φορές βρισκόμαστε σε σχέση ειρηνικέ, αλλά άλλες φορές έχουμε προστριβές και ε, έτσι πολλές φορές πρέπει να ε, δούμε τι γίνεται στην γειτονιά και πρέπει επίσης να δούμε τώρα σαν σέλφι, σαν αυτοφωτογράφηση τι γίνεται στην περιοχή. Να πρώτα πρώτα η Συρία. Χάος, τραγωδία, ε, αναστάτωση. Δεν τρέφουν πάρα πολλές ελπίδες προς το παρόν για αυτή την κατάσταση, αλλά χρειάζεται παρόλα αυτά να δούμε το φως στην άκρη του τούνελ. Και προσπαθούμε από την πλευρά μας να δούμε τι θα γίνει με το ανθρωπιστικό χάος. Να μπορέσουμε να φροντίσουμε τις χιλιάδες των σύρων, των τραυματιών του πολέμου και έχουμε οικοδομήσει ένα νοσοκομείο στα σύνορα με την Συρία και κάθε μέρα γιατροί και νοσοκόμες δικοί μας προσπαθούν να ε, σώσουν, να σώσουν ή να βοηθήσουν, ε, να φέρουν κάποια λογική, να φέρουν ε, ε, κάποια φυσιολογικότητα σε, αυτή τη, σε αυτόν τον ωκεανό δυστυχίας. Η Αίγυπτος. Στην Αίγυπτο όπως τα γνωρίζετε έχουμε ένα καθεστώς όπου μετά από πολλά χρόνια εντάσεων εντοπίστηκε ότι το πρόβλημα της Αιγύπτου είναι οι ριζοσπάστες Ισλαμιστές και όχι το Ισραήλ. Έχουν καταλάβει ένα τμήμα της χερσονήσου του Σινά. Προσπαθούμε να φρενάρουμε αυτή την οργάνωση γιατί στόχος τους είμαστε και εμείς. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο είναι δυνατόν όλες τις δυνάμεις που καταπολεμούν το Ισλαμικό κράτος στο Σινά. Ε, πάντως, όλα αυτά ακόμα είναι αβέβαιο το πότε θα τερματιστούν. Πάντως, έχουμε την άλλη μεριά τον Λίβανο. Γνωρίζετε στο Λίβανο πόσο προβληματική είναι η κατάσταση. Και την τελευταία δεκαετία δεν είχαμε κάποια σύγκρουση με τους Λιβανέζους. Το τελευταία φορά είχαμε το 2011, είχαν εμπλακεί σε αυτόν τον ε, πόλεμο και με το Ιράν, αλλά τέλος πάντων ε, άγνωστο πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στη Συρία και πότε ξανά θα αρχίσουν ε, κάποια προβλήματα μεταξύ των Σιητών του Λιβάνου γιατί είχαμε μια σειρά από πυράβλους που βομβάρδιζαν όλο το Ισραήλ και επομένως είναι άγνωστο το τι θα γίνει στο μέλλον. Οπότε το σημαντικό το οποίο σας αφορά και είμαι σίγουρος ότι θα υποβάλλετε μία σειρά ερωτήσεων είναι το Παλαιστινιακό. Η εμπλοκή η διαφορά, η προστριβή που έχουμε με το Ισραήλ. Υπάρχουν δύο σχολές σκέψης αυτή τη στιγμή. Από τη μία μεριά έχουμε την Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ στην ε, Γάζα. Εμείς αποχωρήσαμε από εκεί πριν από 10 χρόνια και ελπίζαμε ότι έτσι θα σηματοδοτήσουμε ένα καινούργιο μέλλον, μια καινούργια εποχή στις σχέσεις των δύο λαών. Ήταν πολύ σημαντική η πρωτοβουλία μας το 2006, πολύ θεραλία. Οπότε και ε, είδαμε τι γίνεται στην Γάζα, τι γίνεται ε, γιατί, γιατί τους δώσαμε ε, τη Γάζα των Παλαιστίνης της Παλαιστινιακής Αρχής και προσπαθήσαμε έτσι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε ούτως ώστε να οικοδομηθεί μια συσύμπτωση σύνταξη των δύο λαών δυστυχώς σύντομα μετά την αποβολή χιλιάδων Ζελινών, είχαμε ε, οικισμούς ε, που χτίστηκαν, η Χαμάς ε, είχε το πάνω χέρι με κάποιο είδους πραξικόπημα. Σκότωσε Παλαιστινίους της Παλαιστινικής Αρχής. Πάρα πολλοί Παλαιστίνοι ξεφύγανε μέσω Ισραήλ και φτάσαν στη Δυτική Όχθη. Αλλά από τότε είχαμε τρεις γύρους με ξεσπάσματα βίας και έγινε δορυφόρος του Ιράν η Γάζα. Έχει τους πιο σύγχρονους πυράβλους. Έχει μια σειρά σειράγκων. Ό,τι όπλο μπορείτε να σκεφτείτε. Δυστυχώς ούτε εκεί μπορούμε να δούμε φως στην άκρη του τούνελ για την κυριαρχία της Γάζα. Και αυτό γιατί έτσι υποβαθμίζεται, άμα βρώνεται η άλλη πλευρά, η πιο ρεαλιστική του Ισραήλ, του μας που είναι κατά της τρομοκρατίας και της βίας και τον πιστεύουμε κάθε φορά που μας μιλεί για προσαρμογή, για προσχώρηση στην διζωνική ε, λύση, στη λύση των δύο κρατών για δύο λαούς. Παλαιστίνη για τους Παλαιστινίους, και το Ισραήλ και τους Ισραηλινούς. Και ότι ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι οι διαπραγματεύσεις. Και από το 2014 σηκώθηκε και αποχώρησε από τραπέζι διαπραγματεύσεων και από τότε ε, τα πράγματα έχουν ε, παγώσει, δεν ξαναγυρίζει στις διαπραγματεύσεις, οπότε όσο δεν μιλάμε θεωρούμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται και ε, έτσι υποφέρουν και δύο πλευρές. Να, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στο Ισραήλ. Έχουμε επίση τι τρομοκρατικέ επιθέσει σχεδόν κάθε μέρα ακόμα και σήμερα κάτι έγινε. Έχουμε αθώου πολίτες που πλήσονται. Ε, αυτό δεν μας οδηγεί πουθενά. Να τα αναλύσουμε αργότερα. Τώρα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με το Ιράν εν τέλει. Ακούσατε το κ. σήμερα το πρωί. Άκουσα τι είπε. και είπε ε, για τον Αχμαντινετζάδ και για το Ισραήλ. ο οποίος ε, είχε αναπτύξει ολόκληρο σεμινάριο για το πώς θα είναι ο κόσμος χωρίς τους σιωνιστές. Οπότε και σήμερα τα ίδια λένε βέβαια χρησιμοποιούν πιο ευγενείς διατυπώσεις, πιο διπλωματικά κείμενα, αλλά τόσο δεν ξέρουμε πού θα πάνε και οι σχέσεις μας με το Ιράν. Η ε, αλήθεια είναι ότι είμαστε κάπως απογοητευμένοι από το πώς και πού κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό τώρα είναι περασμένα, ξεχασμένα, αλλά ε, δεν πρόκειται αυτό να σβηστεί από την ιστορία, την ιστορία του κόσμου, τη δική μας ιστορία. Όλα όσα έγιναν στο Ιράν, το κατά πόσον θα τηρήσει ή όχι συμφωνία, τι θα γίνει 10 χρόνια μετά τη συμφωνία, κατά πόσον το Ιράν θα γυρίσει πίσω ε, στην παραγωγή ε, των πυρηνικών. Αυτό μόνο το μέλλον θα το δείξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου χαρά είμαι εδώ κύριε Πρόεδρε. Και με μεγάλη μου χαρά να απαντήσω τις τυχόν ερωτήσεις. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΚΝΕΣΕΤ, ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Είναι καλή ιδέα να ερχόμαστε σε επαφή με τους συναδέλφους μας, τους βουλευτές του Ισραήλ. Όπως είπα, η χώρα είναι σημαντικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια περιοχή που περνάει πολλές αναταράξεις. Το είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, τη μόνη δημοκρατική χώρα της περιοχής και όπως προανέφερα, επανειλημμένα, είμαστε άδικοι συχνά, υπερβάλλοντας στις επικρίσεις που απευθύνουμε εναντίον σας. Και θεωρώ ανεπαρκή την πρόσφατη απόφαση που ελήφθη που έριξε Ελλάδα στη φωτιά. Δύο ερωτήσεις έχω. Η πρώτη. Αν θα υπάρξει επανασύνδεση των σχέσεων με την Τουρκία. Κάθε φορά που συναντώμαστε με τον πρεσβευτή έθεσα το ίδιο ερώτημα. Πότε θα ξαναρχίσουν οι επαφές με αυτή τη χώρα. Δεύτερον, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα των πυρηνικών με το Ιράν και τη θέση του Συμβουλίου του Ιανουαρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η δισταγμή σας όσον αφορά τη συμφωνία που συνήφθη πέρσι πώς να το πω, δισταγμοί σας έχουν υποχωρήσει. Οι παλαιθεύσεις του Διεθνούς, Διεθνούς Οργανώσεως για την Νομική Ενέργεια σας δημιούργησαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ε, συμφωνία που συνήφθη ή πάντα έχετε μεγάλους δισταγμούς όσον αφορά αυτή την ε, ε, συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος. Επόμενος ε, ο ο συνάδελφος Καν. Ένα μισή έως δύο λεπτά παρακαλώ. Γιατί στη συνέχεια έχουμε τον ε, πρόεδρο της Εκνευρωτικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Κύριε Σκάνε, ευχαριστώ πάρα πολύ και να σας καλωσορίσω και εγώ εδώ. Για το θέμα της Παλαιστίνης. Ξέρουμε τις δυσκολίες ε, τις οποίες περνάει η Μέση Ανατολή και ξέρουμε επίσης ότι το Παλαιστινιακό ήταν ένα από τα πιο παλιά θέματα. Άλυτο Είμαι μέλες της αντιπροσωπείας του GCC και συνομίλησα με πολλούς ανθρώπους. Φυσικά το θέμα της τρομοκρατίας είναι στο επίκεντρο. Ένα από τα θέματα το οποίο προκύπτει από το GCC είναι ότι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα που θα μπορούσαμε να πετύχουμε είναι αν επιλύσουμε το Παλαιστινιακό, αλλά αυτό θα, έχει, θα εμπλέξει και το θέμα των εξτρεμιστών. Το μεγαλύτερο ρόλο θα το παίξει το ρόλο του το, το κράτος του Ισραήλ. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε προκειμένου να υπάρξει ψήφισμα. Εγώ εδώ και δεκαετίες προσπαθώ να οικοδομήσω σχέσεις μεταξύ μουσουλμάνων και Εβραίων στην Βρετανία. Εμείς σίγουρα θα επωφελούμαστε. Δεύτερο θέμα σε ό,τι αφορά τη Συρία. Η κατάσταση είναι δύσκολη στη Συρία και τα μέρα με τη μέρα. Ξέρουμε ποια είναι τα ρωσικά συμφέροντα στην περιοχή. Αλλά οι Ιρανοί τι συμφέροντα έχουν, τι προσπαθούν να πετύχουν. Οι Ιρανοί, ναι, οι Ιρανοί. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνεκα, καλώς ορίζουμε. Σας καλωσορίζουμε και κι εμείς. Είμαστε το ECR και είμαστε μεγάλος φίλος του Ισραήλ γενικά στην ομάδα μας. Δύο ερωτήσει. Καταρχάς, σήμερα το πρωί ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον κύριο Ζαρίφ, και του έθεσα κάποιες ερωτήσεις. Ιδιαίτερως μία ερώτηση για το θέμα του ψηφίσματος 1929 του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε ό,τι αφορά τα, συστήματα, τα βαλιστικά συστήματα, σε ό,τι αφορά και την χρήση πυρηνικών όπλων που απαγορεύεται από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν μου απάντησε στην ερώτησή μου. Θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί λοιπόν σε ό,τι αφορά τις μακροπρόθεσμες προθέσεις του Ιράν, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη τεχνολογία βαλιστικής. Και γιατί χρειάζονται καν τέτοιου μεγάλου βελενικού ε, όπλα ως περιφερειακή δύναμη. Ένα άλλο θέμα πολύ επικίνδυνο για τη Συρία. Ο Πούτιν μου δίδεται η εντύπωση, βομβαρδίζοντας πολίτες ε, στην περιοχή, προσπαθεί όχι μόνο να καταστρέψει τα βασικά προπήρια των ε, ε, επαναστατών του, Ρωσικού, του Συριακού στρατού, αλλά να περιορίσει και την πρόσβαση των πολιτών και να αυξήσει την ε, ροή των προσφύγων για να αποσταθεροποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατά πάσα πιθανότητα και την ε, περίοδο που θα γίνει το δημοψήφισμα στη χώρα μου να προσκαλέσει και ένα Brexit ως αντέδραση. Και αυτό θα είναι δώρο σε όσους θέλουν να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ είναι λοιπόν πολύ δυσίωνη η ατζέντα του Πούτιν. Αλλά η μακροπρόθεσμη ατζέντα έχει να κάνει με την καταστροφή των ε, μη εξτραμιστών, μαχητών και να πρέπει να διαλέξουμε τον Ασάντ, τη Ρωσία και την Άισις από την άλλη και θα πρέπει να κάνουμε την επιλογή μας και επίσης αν αναγκαστούμε να επιλέξουμε τι θα επιλέγατε εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριο Αστροπίτσιου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για μια ανταλλαγή απόψεων η οποία είναι σημαντική. Είναι σημαντικό να ακούμε τα πράγματα από την πρώτη πηγή. Θα ήθελα να σχολιάσω για το Ισραήλ ε, και το ότι είναι μια εύρυθμη ε, δημοκρατία στην περιοχή. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο καλό παράδειγμα το οποίο ελπίζουμε στο μέλλον να ακολουθήσουν και οι γειτονικέ χώρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση. Αντίθετα με κάποιου συναδέλφου μου, δεν είμαι βέβαιο ότι γνωρίζουμε ποια είναι τα συμφέροντα των Ρώσων σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του στην Συρία. Δεν βλέπω κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, αν θέλετε. Η καταστροφή της Συρίας, η καταστροφή της αντιπολίτευσης, η δημιουργία κάτι συγκεκριμένο στην όλη περιοχή. Θα ήθελα να σχολιάσετε σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχει ειλικρινές ε, ενδιαφέρον κάποιων μεγάλων δυνάμεων της Ρωσίας ε, στην ειρηνευτική διαδικασία στη Συρία. Δεν είμαι βέβαιος. Ε, με 1.600 πτήσεις και παραπάνω σε δύο εβδομάδες και με τη... το βομβαρδισμό σχολείων και νοσοκομείων ναι, νομίζω ότι η πιο μεγάλη καταστροφή προκαλεί κανεί ε, και από τον υφιστάμενο πόλεμο. Ήστερα, σε ό,τι φορά θα κράτη του Περσικού κόλπου. Πώς πιστεύετε ότι ο ρόλος τους μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση στη Συρία και αναφέρομαι στην ε, αποστολή, για παράδειγμα, ε, μαχητικών αεροσκαφών από πλευρά της Τουρκίας προσφάτως. Ευχαριστώ. Κύριε Σακοράφα. Κύριε Χάνεγκμπιτ, το κράτο του Ισραήλ δημιουργήθηκε από του νικητέ του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αναγνωρίστηκε από τα, ε, από τα Ηνωμένα Έθνη με το ψήφισμα 147 του 47, με συγκεκριμένα σύνορα βέβαια. Σήμερα οι συνομιλίε που πραγματοποιούνται για την ειρηνευτική διαδικασία με τη συμμετοχή και τη Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπουν τη δημιουργία δύο ανεξάρτητων κρατών στα σύνορα που διαμορφώθηκαν το 1967. Παρόλα αυτά, τον περασμένο μήνα το Ισραήλ επιβεβαίωσε τη συνέχιση των επικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αγνώντα και παραβιάζοντα όπως πάντα τι καταδικαστικέ αποφάσει όλων των διεθνών οργανισμών, ενώ ταυτόχρονα κατέστρεψε έξι χρηματοδοτούμενε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρωπιστικέ δομέ, γιατί όπω υποστήριξε ο κ. Νετανιάχου, κατασκευάστηκαν παράνομα. Ε, επιπλέον, την περασμένη εβδομάδα οι Ισραηλινές αρχέ απαγόρευσαν για μια ακόμη φορά και χωρίς καμιά απολύτως δικαιολογία την, την ε, είσοδο στη Γάζα σε επίσημη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πράγμα που έχει ξαναγίνει όσον αφορά τους Ευρωπαίους βουλευτές, αλλά έγινε η ίδια απαγόρευση και στη Διεθνή Αμυστία, σε διεθνείς παρατηρητές, δημοσιογράφους, ειδικούς συζητητές των Ηνωμένων Εθνών και ανταχώ επιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ρωτώ λοιπόν ευθεώ. Ποια είναι τα σύνορα του κράτους που σήμερα εσείς εκπροσωπείτε εδώ. Δεύτερον, αποδέχεστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί παράνομες ανθρωπιστικές δομές. Τρίτον, με ποια δικαιοδοσία απαγορεύει το κράτος σας την είσοδο στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και τέταρτον, θα μου επιτρέψετε μια προσωπική ερώτηση. Είμαι Ευρωβουλευτής και Παλαιστίνια υπήκος και κατέχω επίσημο Παλαιστινιακό διαβατήριο. Θα σα παρακαλούσα λοιπόν να μου πείτε με αυτό το Παλαιστινιακό διαβατήριο μπορώ να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να μου πείτε αν μπορώ να πάω στο Ισραήλ με αυτό. Ένα λεπτό λέει ο πρόεδρο. και οι Ισραηλοί συνάδελφοι επίση θα ήθελαν να μιλήσουν. Από ένα σημείο και πέρα λοιπόν θα σας διακόπτω για να δώσω και την ευκαιρία στους Ισραηλινούς συναδέλφους να πάρουν το λόγο. No, no, forgotten. Έχασα συγγνώμη. Ο κύριος Κάβο. Δεν, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για πρώτη φορά από όταν εξελέγην άκουσα ότι είναι η μόνη πραγματική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή του Ισραήλ και γι' αυτό το λόγο όλες οι πλευρές του Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι πιο συμφιλιωτικοί όσον αφορά τα σχόλια και την ρητορική του Λοιπόν, σας χαιρετώ κύριε Υπουργέ. Σαν φίλος του Ισραήλ ήταν προνόμιο για μένα και καθήκον να ε, υπογραμμίσω τις αντιφάσεις που προέρχονται από τις θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όπως τη θέση για, τις, ε, για τους καταβλισμούς. Ε, στο Στασβούργο μίλωσε η θυματοδότηση για την Μπετσέλεμ, τη μη κυβερνητική οργάνωση, που θέτουν σε κίνδυνο τους Παλαιστινίους που θέλουν να απολύσουν τις γιές τους στο Ισραήλ. Τι αντίκτυπο έχουν να μπουν τα Ισραηλινά αγαθά στην Παλαιστίνη. Πώς επηρεάζεται η παραγωγή. Αυτοί που στηρίζουν τους Παλαιστινίους στηρίζονται. Αλλά απ' την άλλη έχουμε τη Χαμάς που ζητάει την καταστροφή του Ισραήλ. Άρα είναι επιβλαβές αυτό για ε, ε, το Ισραήλ. Πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν επικλήσει για την εξολόθρευση του Ισραήλ. Η, Γκόλτα η είχε πει, αν οι Άραβε τελικά θα τα όπλα του, δεν υπάρχει πόλεμο. Εάν παρατήσουν τα όπλα του Ισραηλινοί όμω, είχε πει η Γκόλτα Meir, δεν θα υπάρχει πλέον Ισραήλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλώ ορίσατε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μία σύντομη ερώτηση έχω να κάνω Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά κοινά συμφέροντα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. Ένα από τα πιο προφανή τέτοια συμφέροντα σήμερα είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το Ισραήλ περιτριγυρίζεται από τρομοκρατικές οργανώσεις, σε Χαμά, στη Γάζη, πολλά στο Λίβανο, Ισλαμικό κράτος στη Συρία, Αλκάιδα στο Σινά και ούτω καθεξής. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την συνεργασία μα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη τρομοκρατία, Τι μπορούμε να διδαχθούμε από τις δικές σα εμπειρίε στον πολύ σημαντικό αυτό κλάδο. Ευχαριστώ. Euh, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ και έχω τρεις ερωτήσεις για σας που είναι σύντομες πρώτα-πρώτα εγώ μεσογειστής δημοκράτης και ήρθε ο κύριος Σιλικπαρό, ένας συναδελφός σας που είχε πολύ σημαντική πρόταση για τις ε, Παλαιστινιο-Ισραηλινές σχέσεις. Θα ήθελε ο κύριος Μπάρ να παράσχει αναβαθμισμένα μέσα και δυνατότητες στην Παλαιστινιακή Αρχή, ούτως ώστε να γίνουν ε, αξιόπιστος συνομιλητής για την ειρήνη. Δεύτερον, η Γαλλία ανέλαβε μια πρωτοβουλία ούτως ώστε στον ΟΗΕ να συγκροτηθεί ένα διευρυμένο κουαρτέτο με Άραβες, Ισραηλινούς και όποιον άλλο θέλει να υποστήριξει την υπόθεση αυτή. Τι λέτε. Επίσης, ο Μωάμεθο Έκτος, ο βασιλεύς του Μαροκού, ε, κανούν σε μια συνάντηση μεταξύ Μαχμούτα Μπά και Βενιαμίν Νετανιάχου, ώστε να δοθεί μια όθηση στην ειρηνική διαδικασία μέσω του Σαμπέν Σιτρί, του επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Μαροκινών Ιουδαίων. Τι λέτε γι' αυτό. Ο κ. Ματοζιόλ, ο οποίος είναι ο πρώτος αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ τους βουλευτές της Κνεσέτ που ήρθαν εδώ για να συνομιλήσουν με το κοινοβούλιο μας. Κάθε μέρα η Ευρώπη ακούγονται πράξεις αντισημιτισμού στην Ευρώπη. Υπάρχει γενική διαφορία της Ευρώπης. Εδώ και μερικούς μήνες στην Guardian είδαμε δημοσιεύεται με ανακοίνωση 300 πανεπιστημιακών Αγγλικών που καλούσαν να γίνει ένα μποϊκοτάζ κατά των Ισραηλινών πανεπιστημίων. Η σουηδική κυβέρνηση εδώ και μερικές εβδομάδες χρηματοδότησε για 104.000 ευρώ ένα βιβλιάριο και ονομαζόταν Επικοκρατία και Απατχάιτ και ε, κατηγορούσε για εθνοκάθαση το Ισραήλ. Καθημερινά στην Ευρώπη διαπράττονται πράξεις αντισημιτισμού στη γενική αδιαφορία που επικρατεί, χωρίς να καταλάβουν ότι ο αντισημιτισμός είναι η μητέρα κάθε μορφής τρομοκρατίας. Διερωτώ με και ρωτώ. Πώς αλλάζει η αντίληψη για την Ευρώπη στο Ισραήλ κάθε φορά που διαβάζουν στο Ισραήλ τέτοιες πράξεις, ε, για τέτοιες πράξεις αντισημιτισμού ή μποϊκοτάζ ε, εναντίον του Ισραήλ. Ευχαριστώ. Ο κ. Βάικλ, είναι ιδιαίτερη ευκαιρία να μπορούμε να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και σας ε, συγχαίρω και για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Νομίζω ότι είναι πολύ περιορισμένες οι συναντήσεις μας και οι άμεσες επαφές μεταξύ των ε, βουλευτών της Κνεσέτ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, προκύπτουν πολλές ε, παρανοήσεις ό,τι αφορά τις προθέσεις μας. Ε, είμαστε επικριτικοί για κάποια στοιχεία. Ελπίζω να κατανοείτε ότι πιο πολλοί εξημών είμαστε φίλοι της χώρας σας ότι... και ανησυχούμε για την ασφάλεια της χώρας σας. Και γι' αυτό τον λόγο συχνά εμπλεκόμαστε σε ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να μην σας αρέσουν. Τέτοιου είδους λοιπόν ερωτήματα θα ήθελα να σας θέσω. Κατανοώ ότι ήσασταν και υπουργός, ε, έχετε διατηλέσει και υπουργό δικαιοσύνης ε, στη χώρα σας. 6.666 ε, φυλακισμένους έχετε στη χώρα σας σε διάφορες θέσεις, μεταξύ των οποίων 700 ανήλικοι, παιδιά. 580 είναι οι διοικητικά κρατούμενοι. Μιλώντας, συνομιλώντας με τα άτομα τα οποία μας επισκέπτονται από λιγότερο δημοκρατικές χώρες σε σχέση με το Ισραήλ, ρωτάμε και θέτουμε θέμα για τρεις, τέσσερις, δέκα κρατούμενους. Εσείς έχετε 6.000. Τι θα κάνετε με τα 6.000 αυτά άτομα. Τι περιμένετε από τα 700 αυτά παιδιά που κρατούνται σε φυλακές. Πώς μπορούν να αναπτυχθούν και να καταστούν φίλοι της χώρας σας, φίλοι των παιδιών σας. Ευχαριστώ πολύ. Thank ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε για την ε, παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σας εδώ. Εγώ είμαι από την ομάδα των Πρασίνων. Είμαστε φίλοι της ειρήνης στη Μέση Ανατολή γενικά. Ήθελα να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα για τη Συρία. Το Δεκέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου, ακούσαμε τι έγινε με τον Πρωθυπουργό Νετανιάου και τον Πρόεδρο Πούτιν γίνεται κάποια συζήτηση χαμηλότερο επίπεδο με την Ρωσία για τη Συρία και ποια είναι τα θέματα αυτά, αν μπορείτε βέβαια να αποκαλύψετε κάποια εξ αυτών. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη σύμπτωση. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Μεγάλη σύμπτωση που συναντιόμαστε. Μόλις επέστρεψα, ξέρετε. Σαν μέρος αντιπροσωπείας για την Παλαιστίνη. Επέστρεψα λοιπόν από τα κατεχόμενα εδάφη. Τεπεσκέφθην για πέντε μέρες την περασμένη εβδομάδα. Και μου έλειπε η ζαλινή φωνή. Δεν μιλήσαμε τους ζαλινούς. Εκτός από ΜΚΙΟ. Έχω μία δύο ερωτήσεις. Οι πολιτικοί ηγέτες μας είπαν κάτι. Ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες η Αμάς και η Φατάχ να συνομιλήσουν στην Τόχα και να βρουν κοινό έδαφος. Και τελικά να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση ενότητας. Ποια είναι η θέση του Ισραήλ όσον αφορά μια κυβέρνηση ενότητας. Δεύτερον, από την εμπειρία μας τι διαπιστώσαμε. Ότι 600.000 έπικοι που ζουν στη Δυτική Όχθη ή κατεχόμενα εδάφη όπως αποκαλούνται από την άλλη πλευρά φαίνεται να κατέχουν όλο και περισσότερη γη, να αρπάζουν γη από τους Παλαιστινίους. Και τελικά αυτό που θα οδηγήσει. Τα Παλαιστινικά εδάφη θα χωριστούν από λωρίδες Ισραηλινών επικισμών. Είναι σκόπιμη η πολιτική αυτή του Ισραήλ να μην υπάρχει βιώσιμη επικράτεια ε, Παλαιστινιακή σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο μικροφόνο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας ρωτήσω κάτι για την ε, ε διαδικασία της ειρήνευσης. Γιατί νομίζω ότι αυτά το οποίο μας είπατε ήταν κάτι μανιχαϊστικό, κάπως χρυσώσατε το χάπι, γιατί ε, ε, έχουμε το, τόσα, τόσα πράγματα τα οποία τελικά μας εξωθούν στο να κάνουμε λάθη γιατί το θέμα είναι ότι είναι όλο ένα και ε, περισσότερο επεκτείνονται οι επικισμοί παράνομοι αυτό είναι δικό σας θέμα από την άλλη μεριά θα, ε, πρέπει να δούμε το θέμα τι κάνετε εσείς και ο μεγάλος σας ε, αδελφός που σας βοηθάει δηλαδή είπα αλλά το θέμα δεν είναι μόνο εκεί που έχουν πάει τα πράγματα στραβά είναι το θέμα της δίκης δηλαδή αρνείστε να υπάρχει κράτος δικαίου άλλοι είναι 500 και άλλοι είναι 134 οι οποίοι δεν έχουν δικαιώματα. Ε, όλοι αυτοί είναι στη φυλακή τώρα και μιλάμε για εκατόν τόσα παιδιά ανήλικους που είναι εκεί πέρα. Ε, επίσης, ε, τι, έχουν υποστεί οι δημοσιογράφοι. ασκείται βία εναντίον τους και επίσης είπατε ότι χρησιμοποιείται χημικά, χρησιμοποιείται πυράβλους με κεφαλές χημικές και ε, κάποιος Ισπανός επίσης έχει φωνευτεί που ήταν σε μια βάση του ΟΗΕ στα με το Λίβανο. Οπότε τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται με όλες αυτές τι, λέτε, τις, τις επισκέψεις. Αυτό είναι η εύκολη πρόφαση. Οπότε εσείς ελέγχετε αέρα, θάλασσα και γη εκεί. Επομένως ε, εμείς πώς να περάσουμε εκεί, εμείς οι ευρωβουλευτές δεν μας αφήσαν να περάσουμε. Για πέστε μας τι θα κάνετε αγαπητέ ούτως ώστε να υλοποιήσετε ε, την ειρηνευτική εντολή. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μας αποτρέπουν οι ερωτήσεις με κριτική. Αντιθέτως, αισθανόμαστε ότι είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να σας κάνουμε να μας κατανοήσετε και να κατανοήσουμε και εμείς εσάς. Και όλοι να αντιληφθούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, μην τη Ιδιαίτερα μεταξύ φίλων, αλλά ακόμα και όσοι δεν αισθάνονται φίλοι του Ισραήλ και αυτοί νομίζω έχουν ε, το δικαίωμα να μας ε, προκαλούν με δύσκολες ερωτήσεις. 13 ερωτήσεις. Ε, δεν πρόκειται να αναφερθώ σε κάθε μία εξ αυτών ειδικά, γιατί ακόμα και για ένα λεπτό να μιλήσω για την καθεμία δεν θα βγάλω μακρύ. Τρία ζητήματα όμως ήταν τα βασικά ζητήματα τα οποία έθιξαν οι ερωτήσεις. Ε, το πιο συναισθηματικό, αν θέλετε, το θέμα το παλαιστινιακό. Όλοι μας εδώ πολεμούμε, πολεμήσαμε στο πεδίο μάχης για το Ισραήλ. Τρεις ε, από εμά ήμασταν από πεζοναύτες, ε, από το σώμα αυτών και ο γιος μου πολέμησε στους στον τελευταίο πόλεμο στη Γάζα. Δεν υπάρχει ούτε ένας Ισραηλινός ο οποίος ε, δεν θα ε, έδινε πάρα πολλά για να πετύχει ε, ειρήνη με, το, με την Παλαιστίνη. Με την Ιορδανία και την Αίγυπτο είδαμε ότι αυτές οι χώρες κόστησαν πάρα πολλές χιλιάδες ζώων ε, των Ισραηλινών. Δεκάδες χιλιάδες ήταν οι απώλειες και από πλευρά της Αιγύπτου. Την πρώτη φορά μας που υπήρξε ηγέτης ε, μεταξύ των αραβικών κρατών που μπορεί να κλείσει ειρήνη μαζί μας. Παρατηθήκαμε από τις αρχές ε, της αδιαλαξίας και κάναμε ε, υποχωρήσει. Δώσαμε το Σινά την Ιορδανία για να ζήσουν ε, οι Παλαιστίνοι. Αποδεχτήκαμε πολλές από τις αξιώσεις τους. Εμείς και η Ιορδανία, εμείς και η Αίγυπτος ήδη έχουμε κλείσει δεκαετίες ε, ειρήνη, 40 χρόνια με την Αίγυπτο, 20 χρόνια με την Ιορδανία. Δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω από το να έρθουν σε 20 χρόνια Ισραηλινοί να σας πούν ε, ότι κοιτάξτε έχουμε ήδη 20 χρόνια ειρήνης με, την, με το Ισραήλ. το όνειρο αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο οι Ισραηλινοί ή οι Παλαιστίνοι που πληρώνουν με αίμα το τραγικό αυτό το τίμημα, αλλά και εμείς οι ίδιοι, όχι μόνο με τις ζωές μας, αλλά κάθε μέρα, κάθε μέρα επικρατεί φόβος. Αίσθημα ανασφάλειας Ξέρετε τι συμβαίνει αν κάθε μέρα κάποιος ε, δολοφονείται, πέφτει θύμα ε, βομβιστικής ενέργειας. Όχι μόνο αυτός που πεθαίνει, αλλά και τα 8 εκατομμύρια Ισραηλινοί αντιλαμβάνονται ότι αύριο μπορεί να είναι οι ίδια τροφός τους, ο γιος τους. Ο μοναδικός τρόπος λοιπόν να το πετύχουμε είναι ο τρόπος που πετύχαμε και με τον Βασιλέ ε, Χουσέιν της Ιρδανίας και τον Ασάτ της Αιγύπτου να θέσουμε όλες τις απογοητεύσεις μας, όλες τις συγχύσεις μας, όλα τα ζητήματα ε, και να βρούμε ένα κοινό παρανομαστή και να συμβιβαστούμε. Το συμβιβασμό που περιμένουμε από την Παλαιστίνη έως τώρα οι Παλαιστινοί πρόσφυγες δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να πούν ότι θα γυρίσουν κάποια στιγμή στο Ισραήλ. Δεν το επιτρέπουν. Οι ηγέτες ε, στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο ε, πλήρωσαν το απότατο ε, τίμημα για να κερδίσουν την ειρήνη. Με τη ζωή τους το πλήρωσαν. Τη δικαίωμα της επιστροφής που το... η σημασία είναι το τέλος του Ισραήλ όταν ε, θα αντιληφθούν ότι αυτό το όνειρο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, να επιστρέψουν στο Χαϊφά κτλ. Και, οι φίλοι μας από την αριστερά δεν μπορούν να αποτεχθούν το όνειρο του να επιστραφούν και να επανέλθουν οι Παλαιστίνοι σε άλλες περιοχές. Όλα τα υπόλοιπα ζητήματα είναι τεχνική φύσεως. Πού θα μπουν τα σύνορα, πού θα επιτρέπονται επικισμοί και ποια τμήματα θα συμπεριληφθούν, ε, ποια τμήματα θα ανταλλαχθούν, πώς θα διερθεί η Ιερουσαλήμ, ε, τι τμήμα θα πάει στην Παλαιστίνη, τι ε, τμήμα θα πάει στο Ισραήλ χωρίς να διχαστεί και πάλι η ιερή αυτή η πόλη όπως το Βερολίνι. Όλα αυτά θα λυθούν. Το βασικό ζήτημα είναι για τους Παλαιστινίους. Αυτό που λέμε, αυτό που λέμε ότι ποτέ δεν θα επιτρέψουμε στους Παλαιστινίους να πάνε στα σύνορα πριν από το 67. Κανείς Ισραηλινός δεν θα το αποδεχτεί αυτό. Αυτό είναι ο μεγάλος συμβιβασμός που πρέπει να δεχτούν. Και αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κόσμος, όλος, μας επιτρέψει να πείσουμε τους Παλαιστινίους ότι θα πρέπει να κάνουν αυτή τη μεγάλη υποχώρηση, ότι το όνειρο θα πρέπει να το καταλήψουν κι εγώ, κι εγώ. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι δύο μαχητών που πολέμησαν την κατοχή των ε, Βρετανών ε, το... και φυλακίστηκαν, ε, καταπολέμησαν την Βρετανία και μετά εγκατέλειψαν την ιδέα αυτή με την οποία μεγάλωσε ότι το Ισραήλ δεν είναι μόνο το μικρό Ισραήλ, αλλά και το ευρύ Ισραήλ, Μπασάν, Κοράν, Μογάμ και Ντιλάντ, Ιουδαία και το καθεξής. Το εγκατέλειψαν το όνειρο αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε σε εκατομμύρια ε, οι Παλαιστινίους και η Ιουδία και η Σαμαρία. Θα αποφασιστεί που θα μπουν τα σύνορα, πώς θα τοποθετηθούν τα σύνορα βάσει των αρχών της ασφάλειας. Αλλά το βασικό ζήτημα είναι να κάτσουν μαζί μας και να μας πείσουν ότι θέλουν να ζήσουν ειρηνικά μαζί μας. Αυτό είναι το βασικό. Αν το πετύχουμε αυτό θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε αντί κάθε φορά να τους λέμε ότι βάζοντας επισήμανση και ετικέτες στα Ισραηλινά προϊόντα και με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα τους βοηθήσετε να πετύχουν το, το Παλαιστινιακό κράτος και όχι να κάτσουν μαζί μας να συζητήσουν και να κάνουν υποχωρήσεις. Αυτό, αυτό και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι ηγέτες σας αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, ότι όχι μόνο να συμβάλλετε στην ειρηνική διαδικασία, αλλά φέρετε και κίνητρα να κάτσουν να πετύχουν τον ειρήνη μαζί μας. Έχει αυτή λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου. Έχουμε ένα γιατί τον μας, ο οποίο το κατανοεί αυτό. Δεν είναι ενδεχομένω όσο δυνατό ε, όσο θα έπρεπε. Αυτό ισχύει και για του δικού μα ηγέτε. Αλλά οι ηγέτε θα πρέπει να κάτσουν μαζί και να, κάνουν, να πάρουν αποφάσει. Και τότε θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στο διαβητήριό σα και να πάτε οπουδήποτε στο Ισραήλ. Και θα μπορέσουμε και εμεί να σταματήσουμε να φυλακίζουμε παιδιά. Γιατί αυτά δεν είναι παιδιά, σε εισαγωγικά. Είναι παιδιά τα οποία σε κάποιε περιπτώσει δυστυχώ προσπαθούν να σκοτώσουν Ισραηλινούς πολίτες. Είτε είναι παιδί, είτε δεν δεν έχει σημασία. Αν σκοτώνει Ισραηλινό ή βάζει βόμβες ή μαχαιρώνει, δεν μπορούμε απλά να το αφήσουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να κάτσουμε στο τραπέζι και να κάτσουμε με τους ξαδέρφους μας, τους Παλαιστινίους και να πάρουμε αποφάσεις για την κοινή μας ζωή. Και έτσι μπορεί να είναι ε, πολύ καλή η συνεργασία Παλαιστίνης και Ισραήλ, για το Ιράν. Επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο. Το βασικό ζήτημα, δεν θέλω να επισέλθω στι λεπτομέρειε του JPC, θεωρούμε ότι δεν είναι καλή η συμφωνία, αλλά τώρα είναι η πρόκληση για μας και για σας και για τη ΣΥΠΑ και για όλο τον κόσμο να είμαστε πολύ ισχυροί για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε παραβίαση, παραβίαση τέτοια ε, ε, συμφωνίας. Γιατί θα μας προκαλέσουν και θα μας ε, ε, δοκιμάσουν. Είναι εξαιρετική σε αυτό η Ιρανοί. Αυτοί θα το πούν ερμηνεία, αλλά θα είναι παραβίαση. Να θέσουμε λοιπόν ένα όριο, να είμαστε ενωμένοι, να μιλήσουμε με μια ενωμένη φωνή για να αναγκαστούν να τηρήσουν το λόγο τους. Και τελευταία μου λέξη για τη Ρωσία και τη Συρία. Η Συρία θα ήθελα, αν ακούγονταν η φωνή μου, να φύγει ο Ασάντ είναι υπεύθυνο για το θάνατο 450.000 ανθρώπων. Η μισή του χώρα έχει εκδιωχθεί από τα σπίτια του. Είναι πρόσφυγε μέσα στη χώρα του την ίδια και σε άλλε χώρε. Εγώ πιστεύω και η όραμά μου είναι ότι η δημοκρατική Συρία με τι νέε δυνάμει που μετά από τόσα χρόνια καταπίεση, θέλουν και πάλι να αναδειχθούν και να ελέγξουν τη ζωή του, θα αποτελούσουν το τέλος του Ιράν, της Χισμπολά και άλλων δυνάμεων που προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον κόσμο και τη Συρία. Και θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω που μας φιλοξενείτε και εμένα και την αντιπροσωπεία μου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much for this interesting debate. Ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα αυτή τη συζήτηση και πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις αυτέ την επόμενη φορά να οργανώσουμε τη συζήτηση με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρουν τον λόγο και οι συνάδελφοι από την Κνεσέτ. Ας το οργανώσουμε λοιπόν την επόμενη φορά λίγο καλύτερα τα πράγματα, να δικό μου σφάλμα. Και πιστεύω ότι τέτοια ανταλλαγή απόψεων είναι ύψης της σημασίας για μας. Και με χαρά μας θα ξαναλθούμε κι εμείς. Και σας απειλούμε, μπορεί να έρθουμε κι εμείς στη χώρα σας. Ladies and gentlemen, please take your seat. Καθίστε παρακαλώ κυρίες και κύριοι. I now have the great pleasure. Με μεγάλη μου χαρά. Mr. Καλώζω τον κύριο Λίκερτοφ, πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ. Σας συναντήσαμε περασμένο Νοέμβριο εις Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη όταν σας επισκέφθημε στη Γενική Συνέλευση. Με τα χαρά συνεχίζουμε την καρποφόρα ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε εμεί την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιουργήσετε εσεί για μα. Όπω ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τα μάλα των ΟΗΕ. Είναι χρήσιμη πλατφόρμα για τη μετώπιση παγκοσμίων προβλημάτων, όπω βλέπουμε και τώρα. Το Ευρωκοινοβούλιο υποστηρίζει πιο επιφανή ε, ρόλο ε, στην περιφερειακή εκπροσώπηση όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση εντός του ΟΗΕ. Η βελτιωμένη θέση παρατηρητού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είχε θετικά αποτελέσματα, προωθεί την συνένεση, βοηθά το συντονισμό της πολιτικής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εντός της Γενικής Συνελεύσεως και εντός των Ηνωμένων Εθνών αυτών κάθε αυτών. Οι τρει θεματικέ συζητήσει ψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση όνται υπό την ηγεσία σα του επόμενου μήνε αντικατοπτρίζει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που εστιάζεται επί της επιτεύξεως βιωσίμου αναπτύξεως, ειρήνη, ασφάλεια και κυρίως τις επιχειρήσεις του ΟΗΕ υποστηρίζει του ΟΗΕ. Την προάσπιση θέση των γυναικών και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια του ΟΗΕ είναι κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξη. Έχουμε ελάχιστο στη διάθεσή μα. Χωρί να χρονοτριβώ, θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Πόγκα, στον οποίο δίνω αμέσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπροκ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εξοχότητά του, του για που παίρνει το λόγο ενώπιον δύο επιτροπών σήμερα. Να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος της ε, Προέδρου κυρίας Μακέβαν που δεν μπορεί να, έρθει μαζί, να είμαι μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Η Επιτροπή Ανάπτυξη προφανώς δεν είναι τρεις σημασία της εργασίας για την εφαρμογή των στόχων των αναπτυξιακών, των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων και των δικτών ε, που καταρτίζονται και ελπίζουμε ότι θα παρουσιαστεί τον ε, Μάρτιο στην Οικοσόκ. Η μας επίσης ε, συμβάλλει για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη των βιώσιμων στόχων και τον Σεπτέμβριο στην Σύνοδο του Ηνωμένων Εθνών ε, παρουσιάστηκαν αυτά οι 17 στόχοι και θεσμευόμαστε για να πετύχει αυτή η ατζέντα για το 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη και θα συγχαίρουμε για τις ε, επιλογές σας και για το γεγονός ότι θα υπάρχει συνέχεια για τις επίτευξες των στόχων αυτών τον Απρίλιο. Θα πρέπει να είμαστε ενεργοί και να ορίσουμε πώς οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι θα επηρεάσουν την εξωτερική και ιστορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίσκεψη του αναπληρωτή γραμματέα σε ό,τι αφορά και την ατζέντα για το 2030 που συνομίλησε με διάφορους συναδέλφους και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και η επισκέψη του εδώ στην κοινή αυτή συνάντηση είναι πάρα πολύ ωφέλιμη για να δώσει και ένα νέο κίνητρο, μια νέα ορμή και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να προασπίσετε αυτή την πολύ φιλόδοξη Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ λοιπόν για το λόγο, για την δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω στους συναδέλφους μου τους Ευρωβουλευτές. Μεγάλη τιμή που μιλώ σε εσάς. Σαν πρώτος δανός πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσης του ΟΗΕ. Ποια ήταν η εμπειρία μου το πρώτο ήμιση ενεστώτος έτους ως πρόεδρος Πολλές αντιφάσεις αντιμετώπισα και αντιμετωπίζουμε στον κόσμο. Λάβαμε μεγάλες αποφάσεις. Σημαντικές αποφάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για το κλίμα. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο κόσμος οπισθοχωρεί. Ξεσπούν περισσότερες συγκρούσεις Έχουμε ανθρωπιστικές καταστροφές, κύματα προσφύγων που αντιμετωπίζει και η Ευρώπη και που καταφθάνουν στους ακτές μας. Έχουμε θετικές πτυχές και αρνητικές. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ηνωμένα Έθνη έχουμε κοινέ αξίες και κοινή μοίρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό ο ΙΕ έχει ευκαιρίες και είναι ευκαιρίες αυτές και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που αποφασίσαμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το θεματολόγιο για το, μέχρι το 2030 ήταν κάτι επαναστατικό. Θέλουμε να ακολουθήσουμε νέο δρόμο. Ομόφωνα αποφάσισαν 193 χώρες Θέλουμε να αλλάξουμε το πλανήτη και να προωθήσουμε την ειρήνη και την ευημερία. Συλλογικά συμφωνήσαμε. Θεωρούμε ότι απαιτείται αλλαγή. Απαιτείται μεταμόρφωση του συστήματος του οικονομικού, του κοινωνικού και του συστήματος διακυβέρνησης. Ένα τμήμα της μεταμόρφωσης λεπτομερώς αναφέρει τη Συμφωνία για το Κλίμα των Παρισίων ήταν μεγάλο ποιοτικό άλμα αυτό στο θέμα αυτό που είναι υπαρξιακή φύσεως για όλους. Οι συμφωνίες λοιπόν για το κλίμα δείχνουν πόσο σημαντική είναι η θέση του ΟΗΕ και δείχνει και την αλεξάρτηση που έχουμε και σε σχέση με τους αναψυχικούς στόχους που θέτουμε. Αν θέλουμε οι συμφωνίες να καταλήξουν κάπου, χρειάζεται δράση τώρα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ορμή την περσινή, να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια που δημιουργούν οι συμφωνίες σε απτές κινήσεις και δράσεις και στην Ευρώπη και διεθνώς. Ξεκινάμε από μια στέρεη βάση. Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας βοήθησαν να πετύχουμε θαυμάσιες βελτιώσεις όσον αφορά τις εξελίξεις και αποδεικνύει ότι αν ενδιαφερθεί η κοινωνία και είναι ενωμένη έναντι κοινών στόχων μπορεί να πετύχει πολλά. Η αλληλεγγύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσουμε του αντιστοιχικού στόχου ήταν κρισίμου σημασία και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Τώρα, όσον αφορά την αλλαγή, όσον αφορά την οικονομία που θα είναι ανθεκτική όσον αφορά τι αλλαγέ του κλίματο και θα χρησιμοποιεί ελάχιστα τον άνθρακα σαν ενεργειακή πηγή είναι κάτι που μπορεί να προωθηθεί από την κοινωνία των πολιτών, τις εταιρείε, τις πόλεις, δήμους κλπ. Θα πρέπει τώρα να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Θέλουμε βιώσιμη παγκόσμια υποδομή για τα επόμενα 15 χρόνια. Θα χρειαστούν τρισεκατομμύρια δολάρια που θα επενδυθούν. Να επενδυθούν σωστά για βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξη. Τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών θα πρέπει να προωθηθούν. Χρειάζεται να αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα. Να εκριζώσουμε την ακραία φτώχεια, να μειωθούν οι ανισότητες. Η φοραποφυγή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί γι' αυτό και θα πρέπει να δοθεί αναπτυξιακή βοήθεια στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και να αυξηθεί. Θέλουμε ειρηνικές κοινωνίες. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον αποκλεισμό, να προστατεύσουμε τα πολιτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των πολιτών και θα πρέπει να δημιουργηθούν θεσμοί οι οποίοι να, είναι, να συμπεριλαμβάνουν τους πάντες και να τους καλύπτουν. Η μεταμόρφωση δεν θα λάβει χώρα μόνο από τη δράση των κυβερνήσεων. Τεράστιο μερίδιο των επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια και σχετικές υποδομές θα πρέπει να προέλθει από ιδιωτικές πηγές, όπως επιχειρήσεις, ε, κεφαλουχικούς επενδυτές και διάφορα ταμεία. Και γι' αυτό οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο για τις αγορές και φορολογικό πλαίσιο, Ούτω ώστε οι πράσινε επενδύσει να είναι ασφαλέστερες, να είναι οι καλύτερες επενδύσεις, όχι μόνο για την ανθρωπότητα, αλλά και για τι επιχειρήσει εδώ και τώρα. Πολλά μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό. Εγώ από τη θέση μου θα κάνω ό,τι μπορώ. Και θα χρησιμοποιήσουμε το σύστημα το ΙΕ για να προχωρήσουμε. Και ταχύτερα από ό,τι κάναμε πριν από 15 χρόνια όταν ξεκινήσαμε και θέσαμε τους στόχους της χιλιετίας. Υπάρχουν αντιφάσεις όπως ανέφερα πριν από λίγο. Είναι τέτοιες και τελικά λόγω αντιφάσεων και αντικρουωμένων αποφάσεων αντιμετωπίζουμε παγκόσμια κρίση άκρος ανησυχητική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση. Αντιμετωπίζουμε δύο εξτρεμισμό που οδήγησε στη σφαγή αθώων, αμάχων σε όλο τον κόσμο. Αντιμετωπίζουμε και τη διάδοση όπλων όλων των ειδών και αναδύονται νέες απειλές στον κυβερνοχώρο και από παγκόσμιες, σε παγκοσμίων βελίας επιδημίας. Βεβαίως, οι συγκρούσεις κυρίως στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική δημιουργούν μιζέρια, θάνατο, καταστροφή και πόνο για εκατομμύρια. Πολλά θέματα λοιπόν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ΙΕ και το πολυμερές σύστημα εν γέννη δεν πέτυχαν τους στόχους τους γενικά. Ναι, υπάρχουν παραδείγματα όπου η πολυμερής προσέγγιση προστατεύει και τους ανθρώπους και την ειρήνη, εν γέννη όμως δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που πετυχαίνουμε τώρα. Ας σκεφτούμε τη σύγκρουση στη Συρία, όταν αναφέρουμε τα προβλήματα, σίγουρα υπάρχουν χώρες που έχουν μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά η παρούσα κατάσταση δείχνει τα τεράστια ελλείμματα τη συλλογική προσεγγίσεω όσον αφορά την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Δείχνει ότι είμαστε ανίκανοι να προλείψουμε την κλιμάκωση εντάσσεων και να καταλήξουμε συγκρούσει, να προστατεύουμε του αμάχου στι συγκρούσει και να διευκολύνουμε ειρηνικέ πολιτικέ διευθετήσει που χρειάζονται τόσο πολύ. Δείχνει και ανικανότητα να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε μια ανθρωπιστική απάντηση στα προβλήματα. Χιλιάδες πολίτες στη Συρία υποφέρουν από τις πρόσφατες κλιμακώσεις των βομβαρδισμών και των βιοπραγιών. Η βασική ανθρωπιστική βοήθεια εξακολουθεί να μην μπορεί να φτάσει σε εκείνους που τη χρειάζονται και πεθαίνουν άνθρωποι καθημερινά προσπαθώντας να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο στην Ευρώπη και έχουμε εκατομμύρια α, πρόσφυγες που μένουν άστεγοι. Σε αυτό το πλαίσιο είναι κρισίμου σημασία να χρησιμοποιούμε τη Σύνοδο Κορυφής για την Ανθρωπιστική Βοήθεια, που τη συζήτηση θα γίνει τον Ιούλιο υπό την Προεδρία μου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ανθρωπιστικά <coughs> θέματα. Και 19 Σεπτεμβρίου τελικά έχουμε Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά τη Γενική Συνέψη του ΟΗΕ του Φθινοπόρου που θα συζητηθούν τα προβλήματα των μεταναστών, των προσφύγων. Πρέπει να βρούμε πιο αξιόπιστες λύσεις και βιώσιμες λύσεις στην παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση. Τι σημαίνει αυτό. Πολλά περισσότερα χρήματα και στις περιοχές όπου εκτοπιστέντες και οι πρόσφυγες ούτως ώστε να παραμένουν εκεί και να μην έρχονται κατακύματα στην Ευρώπη και να πετύχουμε καλύτερες συμφωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο και με την κατάσταση. Ήρθε η ώρα να προωθήσουμε τις βασικές προδιαγραφές και αρχές που συμφωνήσαμε γενικώ για να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους στον κόσμο, να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προστατεύσουμε τους πρόσφυγες και χρειάζεται μια Ευρώπη η οποία είναι πρόθυμη να ηγηθεί για να τα πετύχουμε όλα αυτά. Αυτά χρειάζεται ο κόσμος. Η παρούσα κρίση των προσφύγων είναι άνευ προηγουμένου σε κλίμακα. Δημιουργεί προβλήματα σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης και δημιούργησε φόβο και πανικό σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσε και σε πολλά ε, τμήματα του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Η ανικανότητά μας να βρούμε λύσεις υπονομεύει και θέτει σε κίνδυνο ζωές και θέτει, ε, δημιουργεί εντάσεις στους δεσμούς που συνένωσαν και δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς υπάρχει κακυποψία μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ πληθυσμών. Μεγάλη καχυποψία. Αλλά πραγματικά ελπίζω ότι τώρα οι ηγέτες μας και αυτό το μεγάλο κοινοβούλιο θα βρουν τρόπους να ανακαλύψουν ξανά τις αξίες που μας ενώνουν, μας ένωσαν τα τελευταία 60-70 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, γιορτάζει την 70η επέτειο ο ΙΕ και πρέπει να αλλάξει για να ανταποκριθεί στα παρόντα προβλήματα. Σαν πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως, στις συζητήσεις τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούλιο θα ζητήσω ως πρόεδρος τα κράτη-μέλη και άλλους να σκεφτούν, να δουν τι χρειάζεται να αλλάξουμε για να βελτιώσουμε την εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί την ειρήνη και την ασφάλεια ο ΙΕ, να βελτιώσει τη δυνατότητα που έχει και να βελτιώσει τη δυνατότητα του ΙΕ να προστατεύει τους αμάχους και να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ό,τι αλλάξει θα είναι στο επίκεντρο της εντολής που θα δοθεί στον επόμενο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος θα διοριστεί αργότερα φέτος. Εκείνη, νομίζω, και χρειαζόμασταν εδώ και καιρό μια γυναίκα γενική γραμματέα πρέπει να βοηθήσει τον ΟΗΕ να ανανεωθεί. Του χρόνου για πρώτη φορά η Γενική Συνέλευση θα έχει πιο επιφανή ρόλο όσον αφορά την επιλογή και το διορισμό. Για φέτος πρώτη φορά έχετε πιο επιφανή ρόλο όσον αφορά το διορισμό. Και τους επόμενους μήνες θα συγκαλέσω σε επίσημο διάλογο τους υποψηφίους και όλα τα μέλη του ΟΗΕ για να αυξήσουμε τη διαφάνεια για την όλη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και για να βελτιώσουμε τις δυνατότητες να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσον αφορά τον υποψήφιο που θα ηγηθεί των Ηνωμένων Εθνών τα επόμενα χρόνια. Αυτά είναι κάποια τα ζητήματα που απασχολούν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά θα ήθελα να κλείσω με ένα μήνυμα εκ βάθους καρδίας, σαν πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Δανίας και σαν υπερήφανος Ευρωπαίος πολίτης. Τι θέλω να πω. Από τη θέση μου τη σημερινή βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά εξακολουθεί να παίζει βασικό ρόλο στη διεθνή κοινότητα των εθνών, αλλά οι παρούσες εντάσεις και διαιρέσεις μπορούν να υπονομεύσουν τη φωνή της, τη φήμη της και κατ' επέκταση την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο η ισχυρή ενωμένη Ευρώπη που εμένει στις βασικές αξίες μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Γι' αυτό πραγματικά ελπίζω ότι όλοι σας θα συνεργαστείτε μαζί μας στον ΟΗΕ για να βοηθήσουμε να επιφέρουμε την Ένωση της Ευρώπης για μία ακόμη φορά και να προωθήσουμε την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας απευθυνθώ σήμερα. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ, ιδίω για την αποστροφή της ομιλίας, γιατί ουδέποτε δεν έχουμε διατρέξει μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι τώρα αυτές τις μέρες ότι διακυβεύονται όλα όσα πετύχαμε τελευταία κονταετία, λέει ο πρόεδρος, γιατί θα πρέπει να βρούμε το θάρρος και συσπηρωμένοι να αναζητήσουμε λύσεις. Σας ευχαριστούμε. Όμως, θα ήθελα να σας ζητήσω να τηρήσουμε ενό λεπτού σιγή γιατί έμαθα ότι ο πρώην Γενικός Γραμματέα Μπούτρος Μπούτρος Γκάλη απεδίωσε Παρακαλώ ενό λεπτού σιγή. Thank you very much. The floor has no Ο Πρόεδρος και τώρα το λόγο κύριος Μπρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι, εδώ κάθομαι. Στο δεξιά σας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που είσαστε μαζί μας. Είναι πραγματικά χαρά μας που σας ε, υποδεχόμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ και για την παρέμβασή σας. Θα ήθελα να σας πω καταρχάς ότι εδώ στις κοινοβουλευτικές μας εργασίες διαρκώς υποστηρίζουμε την ε, ιδέα της ε, αναθεώρησης των Εθνών και της ε, αναζωπήρωσης του ρόλου της Γενικής Συνέλευσης σε ό,τι αφορά και τον συντονισμό των δράσεων που διεξαγάγει ο Παγκόσμιος Οργανισμός των Εθνών. Πώς τοποθετήσετε λοιπόν για το θέμα αυτό για την ε, ριζική αναθεώρηση του τρόπου εργασία των ΗΕ. Έχουμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, έχουμε και την παρουσία των συναδέλφων και να σας πω ότι είμαι και εισηγητής για την πολιτική συνοχής και την πολιτική ανάπτυξη. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν αν το θέμα αυτό το, στη συνοχή της πολιτικής και της ανάπτυξης ε, συζητιέται στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σε ό,τι αφορά και την εφαρμογή της Ατζέντα 2030. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας λοιπόν εδώ σήμερα. Ο κύριος Κιτσούκ. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε λοιπόν εδώ μαζί μας κύριε Πρόεδρε. Είσαστε από τους κορυφαίους δανούς πολιτικούς και από τους παγκόσμιους ηγέτες που προαγάγουν την οικονομική ανάπτυξη. Στη σημαντική αυτή συνάντηση θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να βρίσκει πιο βιώσιμες λύσεις στα παγκόσμια προβλήματα σεβόμενοι τα οράματα των εκάστοτε λαών. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Λέει ο κύριος εγώ θα ήθελα να υποβάλω την εξή ερώτηση. Όσον αφορά για την Μινούρους, δηλαδή αυτή την ε, αποστολή του 1991 όσον αφορά την ε, Κεχηρία και όσον αφορά το δημοψήφισμα για την Δυτική Σαχάρα και την ε, κατάληψη και κατοχή από πλευρά του Μαροκού έγινε δημοψία. Γιατί εγώ τον Οκτώβριο είχα την τιμή να είμαι σε αυτή την ε, ειδική αποστολή όσον αφορά ε, τον ΟΗΕ στην ε, Νέα Υόρκη και μελετήσαμε, συζητήσαμε τι αυτό. Οπότε σα παρακαλώ, τι θα κάνει ο ΙΕ ούτως ώστε να μπορέσει να βοηθήσει αυτή την, αυτό το δημοψήφισμα που είναι μια εντολή που υπάρχει ε, σε μια από τις ε, τελευταίες απικίες ούτως ώστε να απελευθερωθεί η επικράτεια αυτή από το Μαροκό. Επόμενος, στα γερμανικά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση θα ήθελα να σας θέσω, αν και το αναφέρατε ήδη. Είπατε ότι θέλετε πιο πολύ ε, διαφάνεια για την επιλογή και εκλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Το καλωσορίζω ασφαλώς αυτό. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε πώς μπορεί να διαμορφωθεί η διαδικασία εκλογής. Και μια δεύτερη ερώτηση. Συνομιλήσαμε και με την Τρίτη Επιτροπή σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι ακούσαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα. Και εν ώψη και της μελλοντικής γενικής συνέλευσης θα μπορείτε να μας πείτε τι συζητιέται ακριβώς στους κόλπους της Επιτροπής σας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ και καλώς ορίζω. Καλώς ορίσατε μάλλον στο πιο σημαντικό κοινοβούλιο του κόσμου. Δύο ερωτήσεις καταρχάς σε ό,τι αφορά το θέμα της εκλογής του Γενικού Γραμματέα. Ξέρουμε όλοι ότι τις τελευταίες δεκαετίες η διαδικασία ορισμού του νέου Γενικού Γραμματέα δεν ήταν πολύ διαφανής. Ελπίζουμε λοιπόν αυτή τη φορά να υπάρχει κάπως μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία αυτή. Ποια είναι λοιπόν η άποψή σας. Ο επόμενος Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να είναι από την Ανατολική Ευρώπη. κοιτώντα και από πού προέρχονται οι έω τώρα γενικοί γραμματεί, ή είναι πιο σημαντικό ο επόμενο γενικό γραμματέα να είναι γένο τελικού. Κοιτώντα του υποψηφίου και άλλε γεωγραφικέ ομάδε θα μπορούσαν να προβάλλουν σημαντικού υποψηφίου. Ποια είναι η άποψή σα, και δεύτερη ερώτηση για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όλοι ξέρουμε ότι κάποιοι από τους συναδέλφους ε, έκαναν πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη. σε ό,τι αφορά θέματα γενοκτονιών ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Πόσο έχει προχωρήσει λοιπόν το θέμα αυτό και πιστεύετε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα είναι έτοιμο να περιοριστεί, θα είναι πρόθυμο να περιοριστεί, να αυτοπεριοριστεί σε ό,τι αφορά τη χρήση άρνηση κυρίας Βέτο. Eh, jag skulle στα σουηδικά να σας τα πω, λέει η κυρία Πόρστα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Όσον αφορά το τι κάνετε και στο θεματολόγιο σας, πόσο υψηλά είναι το πρόβλημα των Ρωμά παγκοσμίω. Μιλούμε για 10 εκατομμύρια περιθωριοποιημένοι, δεν έχουν δουλειές, δεν έχουν σχολεία, δεν έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Τι κάνει ο ΙΕ για αυτούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Καστάλτο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Στην Επιτροπή μας, πριν από κάποιους μήνες, συντάξαμε μία έκθεση όσον αφορά για τον ρόλο του ΟΗΕ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι προοπτικές σοβερές και αξιόπιστες υπάρχουν ούτως ώστε να μπορέσετε να μεταρρυθμίσετε τα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είπαμε για το πώς μπορούμε να έχουμε τις περιφερειακές, τα περιφερειακά θεσμικά όργανα στο μέλλον ε, ε, να συμμετάσχουν πέραν των παραδοσιακών πέντε μελών. Τι, τι πιθανότητες υπάρχουν τόσο ώστε κάτι να γίνει. Μήπως θεωρείτε ότι από πολιτικής πλευράς αποκλείεται δεδομένη της συγκυρίας. <clears throat> Καλώ ορίσατε κύριε Κεντροφή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λέγει ο κ. και διότι μου την εντύπωση ότι και στη δική μα επιτροπή μπορεί να βρείτε υποψηφίου για τη θέση του επομένου Γενικού Γραμματέα. Αλλά βέβαια αυτό είναι δουλειά του ΟΗΕ. United Nations is having. σε ποιο βαθμό ο ΟΗΕ έχει ένα σύστημα αποτελεσματικό όσον αφορά ε, κάποιο σύστημα προειδοποίησης όταν δηλαδή ε, ξεσπά κάποια ανθρωπιστική κρίση έχετε ταχεία αντίδραση για αναγνώριση ε, κάποιες κατάστασεις όταν δηλαδή κάτι πάει προς το χειρότερο επίσης κάτι το ρωτάμε και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ε, εκφράζεται στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία φωνή. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σε ευχαριστώ. Λέει ο κύριος Λίκητοφ. Έστω και σε λίγη ώρα θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους. να βρω τη μεταρρύθμιση στον ΟΗΕ, νομίζω ότι αυτό είναι ε, μια κίνηση ενθαρρυντική με μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και έτσι θα πρέπει να γίνει η επιλογή των υποψηφίων για την θέση του επομένου Γενικού γραμματέως. Όλα αυτά θα γίνουν ακριβώς όπως είπαμε. Θα ξεκινήσει η διαδρομή στις 11 Απριλίου και έκαστος των υποψηφίων θα εμφανιστεί στην Γενική Συνέλευση και θα έχουμε μια συνεδρίαση ολομελίας με τον ένα έκαστο εξ αυτών με ερωταπαντήσεις. Θα υπάρχουν επίσης και ερωταπαντήσεις από και προς εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ προηγουμένως. Οπότε αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα. Ε, όπως ξέρετε το Συμβούλιο Ασφαλείας κατεβάζει τις προτάσεις στην ε, Γενική Συνέλευση στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Όμως μέχρι σήμερα τι έχουμε διαπιστώσει ότι οι υποψήφοι ε, συνήθως έχουν μυστικές επαφές με τους πέντε του Συμβουλίου Ασφαλείας και είναι κάπως δύσκολο να συνεχιστεί αυτή η παράδοση εάν τα περισσότερα μέλη ε, του οργανισμού ε, είναι κατά. Και προκύψει ότι θέλουν να υποστηρίξουν ε, τα μέλη ένα συγκεκριμένο υποψήφιο για αυτήν την τόσο σημαντική, την πιο σημαντική θέση που έχουμε στο πολυμερές παγκόσμιο σύστημα. Επίσης δεν έχουμε κάποιες διατάξεις που ορίζουν το αν θα πρέπει να είναι άντρας ή γυναίκα. Είναι ανοιχτή η διαδικασία. δεν ξέρω πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά καταρχήν τώρα θα είναι τα πράγματα πιο δημοκρατικά, πιο διαφανή. Όσον αφορά τη μεταρρυθμίση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Γνωρίζουμε ότι με μια εικοσαετία αυτή η μεταρρύθμιση προχωρά αργά αλλά σταθερά. Δεν είμαι βέβαιος αν μπορώ να υποσχεθώ ότι κατά την μονοετή μου θητεία θα γίνει κάποια μεταρρύθμιση. Αλλά γίνεται συζήτηση υπό την αιγίδα του Λουξεμβουργίου εκπροσώπου για τη μεταρρύθμιση στην Ολομέλεια ή στη Γενική Συνέλευση τέλο πάντων. Οπότε στο μέλλον θα φτάσουμε σε μια τέτοια μεταρρύθμιση κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε κάποια σύνθεση του Συμβουλίου που θα είναι πιο αντιπροσωπευτική. Τώρα όσον αφορά την άρνηση κυρία, το βέτο, υπάρχει και εδώ κάποια σχετική πρωτοβουλία, πρωτοβουλία των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και κυρίως της Γαλλίας και οποιοδήποτε κράτος το οποίο συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας συμμετέχει ή εκλέγεται δεν θα πρέπει να ψηφίζει οποιαδήποτε δράση ε, να καταψήσουμε οποιαδήποτε ενέργεια που οδηγεί σε γενοκτονία. Οπότε αυτό σημαίνει μια καινούργια διοντολογία για τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και ιδίως τα μόνιμα μέλη ε, υποστηρίζονται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης βεβαίως. Αυτό είναι ηθικό το θέμα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ελπίζω ότι όλο ένα και περισσότερο θα είναι μια δηλαδή συντριπτική και όχι απλή πλειοψηφία των κρατών μελών που πρόκειται να υποστηρίξουν αυτό το νέο κώδικα διοντολογίας. Και κατά αυτόν τον τρόπο πρόκειται στο προσκήνιο να ζητηθεί το θέμα για τον περιορισμό ε, της ε, ε, επιλογής του ΒΕΤΟ. Τρόσον φορά τις εξελίξεις για το πολιτικό μας θεματολόγιο μέχρι το 2030 θα πρέπει να υπενθυμίζουμε στις κυβερνήσεις μας και τις ευρωπαϊκές ότι είναι δεσμευμένοι. Έχουν δηλαδή αναλάβει τη δεσμευσή ούτως ώστε το καλοκαίρι αλλά και το φετινό χειμώνα στο Παρίσι να αυξήσουν την αναπτυξιακή βοήθεια προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και έτσι να είναι ευκολότερο το να λιάνουμε τις διαφορές μεταξύ των χωρών. Οπότε είναι απολύτως κατά της αναγκαιότητας το να ελοποιηθούν οι παγκοσμίες συμφωνίες εάν γίνει πίσω γύρισμα στην υπόθεση της ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Είναι και το θέμα των ε, προσφύγων. Δεν θα πρέπει δηλαδή να επικεντρωθεί η ενίσχυση και η βοήθεια μόνο ε, στις άμεσες ανάγκες στα θέματα αυτά των ανθρωπιστικών κρίσεων. και δεν θα πρέπει να κάνουμε πίσω όσον αφορά τις δεσμεύσεις μας για την αναπτυξιακή βοήθεια. Γιατί ανατρέχουν στο απότρο παρελθόν οι υποσχέσεις για την χορήγηση αυτής της βοήθειας. Τώρα, όσον αφορά την Δυτική Σαχάρα, μπορώ απλώς να σας παραπέμψω σε αυτά τα οποία επανειλημμένα έχει αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας όσον αφορά το ότι πρέπει οι εμπλεκόμενοι να συνάψουν κάποια συμφωνία. Όσον αφορά τώρα την Βόρειο Κορέα. έχουμε κατηγορηματικά καταδικάσει τα πυρηνικά πειράματα δια του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και είχαμε κατηγορηματικές διατυπώσεις σε κάποια έκθεση όσον αφορά ε, τα όσα γίνονται εκεί. Και αυτά γίνανε και από πλευρά μια ε, επιτροπή που συνεκρότησε η Γενική Συνέλευση. Στον ΟΗΕ δεν ξέρω τι γίνεται με τους ε, Ρωμά, αλλά βέβαια κατά καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και ε, η διακριτική μεταχείριση εμπίπτουν σε αρμοδιότητες της σχετικής επιτροπής του προγράμματος του ΟΗΕ. Τώρα όσον αφορά τις προειδοποιήσεις, τους συναγερμούς για τις συγκρούσεις, ναι θα πρέπει να βελτιώσουμε αυτό το σύστημα γιατί αυτό όχι μόνο θα πρέπει να, να είναι καμπανάκι για να μας ξυπνάει, αλλά θα πρέπει να επιστρατεύονται και σχετικοί πόροι. Και ακριβώς ε, στο παρελθόν, ακριβώς επειδή υπήρχε κατάσταση ανάγκης απρόβλεπτη, πέρσι κόψαμε στο στο μισό την ενίσχυση μάλλον τις μερίδες φαγητού προς τους ε, πρόσφυγες στην ε, Ιορδανία. Πάντως. Ε, οπωσδήποτε το σύστημα προειδοποίηση επιδέχεται βελτίωση και αυτό και θα κάνουμε. Συμπαθάτε με γιατί δεν έχω χρόνο να μείνω περισσότερο στη συνάντησή μας. Όμως το βλέπω σε μια πολύ σημαντική ευκαιρία που είχα να συμφωνήσω μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ για τις δηλώσεις σας και για τη συζήτηση. Ελπίζω να πετύχετε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την εκλογή του Γενικού Γραμματέα, το ΟΗΕ και για τις μεταρρυθμίσεις του ΟΗΕ. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και νομιμότητα μεγαλύτερη για να βελτιωθεί η αξιοπιστία. Και αυτό χρειαζόμαστε τον ΟΗΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε την υποστήριξή μας. Και να έρθετε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στην έκθεση για την Αλβανία. Και είμαι βέβαιο ότι ο συναδέλφο Φλέκενσταν θα μα ε, ε, ανεβάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο. Και με μεγάλη χαρά, όπω και όλοι οι υπόλοιποι, αναμένω την ε, παρέμβαση του. Άξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη συνάδελφε, το σχέδιο της έκθεσης το έχουμε από τις 26 Ιανουαρίου από την ΑΦΕΤ. Από τον Ιούνιο του 2004 η Αλβανία έχει το καθεστώς υποψηφίας χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει σημαντικές εξέλιξεις και προόδους στου πέντε εντοπισμένου τομεί ω προτεραιότητε, προκειμένου να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσει για την ένταξη. Ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία είναι η μεταρρύθμιση του δικαστικού. Προτεραιότητα στην παρούσα φάση της ε, αλβανικής κυβέρνησης, αλλά και τη ε, αλβανικής αντιπολίτευσης. 90% και παραπάνω των πολιτών της Αλβανίας διατείνονται ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να λάβει η χώρα στην χώρα τους. Περιμένουμε και την τελική γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής της Βενετίας σε ό,τι αφορά τους ε, νόμους που θα περάσουν και όχι μόνο στο πώς θα περάσουν αλλά κυρίως το πώς θα εφαρμοστούν πιο δύσκολο. Ύστερα έχουμε τις άλλες προτεραιότητες, μεταρρύθμιση του, της δημόσιας διοίκησης, καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεμελιωδών, αξιών. Ξέρουμε όλοι ότι χωρίς σωστή μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν να επιτευχθούν οι άλλες στόχοι. Οι άλλες προτεραιότητες, 8 και 9 Φεβρουαρίου Κάναμε συζητήσεις στα Τύρανα με τον συνάδελφο Κούκαν για να ξεκαθαρίσουμε ότι χρειάζεται και συνεργασία πέρα από τα όρια τα κομματικά προκειμένου να τελεσφορήσει και αυτή η προσπάθεια μεταρρύθμισης του δικαστικού σώματο. Και σε ό,τι αφορά το νομοθετικό σκέλος. Ξέρουμε ότι τον Ιόνιο του 2017 έχουμε εκλογές και αν δεν θέλουμε να μπει στην πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση, θα πρέπει να δράσουν άμεσα οι εμπλεκόμενοι φορέ. Από τι συζητήσει μα στα Τύρανα με τον ε, ηγέτη τη αντιπολίτευση τον Πρωθυπουργό, αλλά και με πολλού άλλου φορεί προέκυψε μία περιορισμένη αισιοδοξία τουλάχιστον. Θα παρακολουθήσουμε στενά τη διαδικασία μεταρρύθμισης αυτής. Θα είναι μια διαδικασία εποπτείας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. με τα εφιστάμενα μέσα, με τα εφιστάμενα εργαλεία. Η έκθεση λοιπόν ακολουθεί ένα αισιόδοξο τόνο κυρίως σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση πριν από ένα έτος και σε σύγκριση με την κατάσταση σε άλλες χώρες. Σκοπός είναι να δοθεί κίνητρο στην Αλβανία προκειμένου ε, χωρίς δισταγμό και άμεσα να προχωρήσουν με τις μεταρρυθμίσεις. Η έκθεση αναφέρεται και στις πέντε μεταρρυθμίσεις, πέντε μεταρρυθμίσεων και γνωρίζουμε διάφορα και από την έκθεση πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρουμε ε, ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση καλούνται να περάσουν τις μεταρρυθμίσεις αυτές σε ό,τι αφορά και τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, του Συμβουλίου της Ευρώπης και όλων των υπόλοιπων φορέων. Ελπίζουμε να πετύχει η μεταρρύθμιση του Δημοσίου το 2014 και 2015 ε, είχε ως αποτέλεσμα διάφορα σημαντικά μέτρα, η εφαρμογή των οποίων δεν είναι ιδανική σε κάθε περίπτωση. Η Αλβανία χρειάζεται λοιπόν επαγγελματική και αποτελεσματική διοίκηση για να υπάρξει αυτή η μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και της οργανωμένου εγκλήματος. Έχουν δεσμευτεί μεν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Υπάρχει και ψηφίστηκε μάλιστα και μια στρατηγική κατά της διαφθοράς 2015 2020, αλλά η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων θα πρέπει να εντατικοποιηθεί και υπάρχει μια έλλειψη γιατί δεν γίνονται αρκετέ καταδίκες. Είναι επικοδομητικός εταίρος η Αλβανία στην περιοχή. Είναι ενεργή στο θέμα της περιφερειακής συνεργασίας. Στην Σύνοδο, στο Βερολίνο, στη Βιέννη και η ενεργή συνεργασία με τα εθνικά κράτη-μέλη και με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνονται και από την συζητήσει για το θέμα των προσφύγων, από τις προετοιμασίες που κάνει η χώρα στο θέμα των προσφύγων και από τη στάση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά πρόσφυγες που θέλουν να πάνε στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρονται και πολλά σημεία κριτικής. Οι περιφερειακές εκλογές δεν διοργανώθηκαν με τον τρόπο που θα θέλαμε και συντάξαμε σχετική έκθεση σε ό,τι αφορά επίσης την ανησυχία για τους αλλοδαπούς μαχητές στην Αλβανία. Αφενό δικαιολογείται, αλλά αφετέρου βλέπουμε και τη συνεργασία με τις υπηρεσίες και άλλες οργανώσει της αλλοδαπής και προσπαθούμε να περιορίσουμε το φαινόμενο. Ασκείται και κριτική Υπάρχει και η... το αίτημα να ενισχυθεί η Επιτροπή Σύνδεσης και Συνεργασίας. Οι εσωτερικές διαμάχες στην Αλβανία θα πρέπει να επιληθούν στην προετοιμασία. Και αυτό ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες. Και θα, γίνουν, θα κάνω και εγώ κάποιες ε, προσθήκες σε ό,τι αφορά το θέμα της εκπαίδευσης, το θέμα της, του περιβάλλοντος και της ενέργειας, αλλά προσβλέπω γενικά στα, στη συνεργασία με τους σκιώτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φλέκενστάιν και για την υπόδειξη ότι ο κόσμος ε, με τόσο υψηλά ποσοστά τάσεται κατά της διαφθοράς και υπέρ της μεταρρύθμισης. Αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό αποδεικνύει ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι το εμπόδιο οι πολίτες, αλλά η ενδιάμεση. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να ρευματιστεί η κατάσταση αυτή. Ο κύριος Πρέντα έχει το λόγο εκπρόσωποι των Σκιώδης ηγητή του ΕΛΚ. Ο κ. Χούκαν είναι ο σκιώδης ηγητής, αλλά δεν είναι εδώ μαζί μας. Θα μιλήσω εκ μέρους του συναδέλφου. Όσοι ήδη ανέφερε συγκητής, ο κ. Κούκαν και ο Φλέκενσταν επεσκέφθησαν την Αλβανία μαζί την περασμένη εβδομάδα. Προσπαθούσαν να δούνε ποιε είναι οι πρόσφατες πολιτικέ εξελίξει όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα και την εφαρμογή του νόμου για την αποποινικοποίηση. Ικανοποιήθηκε ο κ. Κούκαν από την επίσκεψη. Βασικό στόχο ε, ήταν να ενθαρρύνει όλου του πολιτικού ηγέτε να πετύχουν πολιτική συνένωση για τι επικείμενε μεταρρυθμίσει. Ο κ. Κούκαν συμφωνεί με τον εισηγητή ότι η Αλβανία έκανε σταθερή πρόοδο να βάσει μεταρρυθμίσει και τι βασικέ προτεραιότητε τον τελευταίο χρόνο και τόνισε ότι η εφαρμογή θα είναι κρισίμου σημασία για περαιτέρω αξιολόγηση. Ο πολιτικός διάλογος και η συνένεση παραμένει το μεγάλο πρόβλημα για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στην Αλβανία. Είναι σημαντικό να τονωθεί ο διάλογος, ώστε να υπάρξει κίνηση προς τη διαδικασία ολοκλήρωσης. Ο νόμος για την αποποινικοποίηση που υθετήθηκε και διαπραγματεύτηκε από το αντικείμενο διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβερνήσεως, πλειοψηφίας και της αντιπολιτεύσεως είναι ένα καλό παράδειγμα πολιτικής συνεργασίας. Η Αλβανία λοιπόν κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ίσως αλλάξουν εις βάθος ε, το χαρακτήρα της χώρας. Σχετικά με αυτό η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα είναι κάτι πολύ περίπλοκο στα διαδικασία Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη-μέλη έχει επενδύσει πολλές προσπάθειες για να βοηθήσει την προετοιμασία των μεταρρυθμίσεων. Όμως θα είναι σημαντικό οι Αλβανοί πολιτικοί να υπομισθούν τις ευθύνες υιοθετώντα και εφαρμόζοντα τη μεταρρυθμίση. Ο κ. Κούκαν συμφωνεί όσον αφορά την αναφορά της Επιτροπής της Βενετίας, των συστάσεων της Επιτροπής Βενετίας για κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. Υπάρχει ευρεία συνένεση μεταξύ Αλβανών πολιτικών ηγετών να ακολουθήσουν τις συστάσεις Επίσης συμφωνεί ο κύριος Κούκαν με την ιδέα να ζητηθεί καλύτερος μηχανισμός ε, εποπτείας για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. Άλλα θέματα υπάρχουν που χρήζουν προσοχής. Η προόδος όσον αφορά την εκλογική διαδικασία και τις εφαρμογές των συστάσεων του ΑΣΕ και μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκηση, καταπολέμηση διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και ελευθερία των ΜΜΕ. Η θετική συνεισφορά της Αλβανίας στην περιφερειακή συνεργασία και η πολιτική βούληση για να βελτιώσει τη σχέση με τη Σερβία είναι κάτι ευπρόσδεκτο από τον συνάδελφο. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι η Αλβανία, η ευθυγραμμίζεται με την ΚΕΠΑ της Ευρωπαϊκής Ενώσης, κοινή πολιτική ασφαλείας, εσωτερική πολιτική. Και τέλος, κάτι εξίσου ο κύριος Κούκαν ευχαριστεί τον εισηγητή διότι ε, προετοίμασε πάρα πολύ καλά αυτή την έκθεση και ο κύριος Φλέγκενστάιν ήταν πολύ ανοιχτός στις συζητήσεις και στην ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Κνούτε για την έκθεση προόδου για την Αλβανία, την Περσινή. Ε, κάναμε συγκεκριμένα βήματα. Η Αλβανία τώρα είναι υποψήφια χώρα, όμως τον τελευταίο χρόνο δεν λάβαμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Επετέφθη πρόοδος σε πέντε κρισίμου σημασία τομείς. Η Αλβανία τώρα έχει στρατηγική για αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης, για μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα κλπ. Πολλά απομένουν να γίνουν όμως για να μεταρρυθμιστεί ο δικαστικός τομέας, για να καταπολεμηθεί η διαφθορά, να καταπολεμηθεί η ανεργία των νέων, να στηριχθεί η ανεξαρτησία των ΜΜΕ, να γίνει επεξεργασία θέσπισης νομοθεσίας και να προωθηθεί πολιτικός διάλογος με συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο κ. Κιουτσούκ πρώτα τα συγχαρητήρια στον κύριο Φλέκινστάιν για τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε για να μπορέσει να συντάξει αυτή την τόσο ε, άρτια έκθεση. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ρόλο της Αλβανίας για την ε, ε, σταθερότητα της περιφέρειας και για τον ρόλο της στην επίλυση του προβλήματος των προσφύγων. Ε, οπότε έχει προσπαθήσει να πληρεί τα κριτήρια για την ένταξη. Ε, έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις στην ε, διοίκηση, έχουν γίνει αποκεντρωτικές κινήσεις και καταπολέμηση της διαφθοράς. Όμως, για τη συνέχεια θα πρέπει να συνεργαστεί η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Να, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα της χώρας, αλλά θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες. Τώρα, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι θετικό πως συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο για την ένταξη στην Ευρώπη. Μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο για τις μεταρρυθμίσεις. Τώρα, όσον αφορά τα λοιπά κριτήρια, τα κριτήρια της Κοπενχάγης, ε, γίνανε προσπάθειες όσον αφορά την αγορά, αλλά ακόμη υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει και σημαντική παραοικονομία. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν θετικά βήματα. Πάντως, είναι εκτεταμένη η διαφθορά και στη δικαιοσύνη και στη διοίκηση. Άρα θα πρέπει η κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες καταπολέμησης. Γιατί η διαφθορά υπονομεύει το κράτος. Είμαι σκιώδης ηγητής για την άλλη. Οπότε σας επισύρω την προσοχή στις θετικές προσπάθειες της κυβέρνησης για την προσπάθεια ελευθεριών και δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι χρειάζεται να ληφθούν μέτρα για όλες τις εθνοτικές ομάδες. Να σταματήσει η περιθωριοποίηση των Ρωμά και των άλλων ευάλωτων. Ευχαριστώ. floor. Now, Mr. Meserich. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ να αρχίσω με ευχαριστίες, με συγχαρητήρια προς ε, τον εισηγητή. Έχω τα εξής τρία σημεία να θα σας πω. Γιατί γενικώ σύμφωνα με το κείμενο. Πρώτα πρώτα είναι βασικό ότι είναι για προστασία των ανηλίκων. Αλλά θα πρέπει να σας προβληματίσει το ότι ο σχετικός επίτροπος δεν καλύπτεται από κονδύλιο του προϋπολογισμού. Άρα, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει από πλευρά ΟΤΑ για μεταρρυθμίσεις. Τι θα γίνει επίσης με την χωροταξία γιατί εκεί οργιάζει η διαφθορά στα Βαλκάνια. Άρα θα πρέπει σε επίπεδο αυτοδιοίκησης εκείνο το θα γίνει. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά θέματα περιβάλλοντας. Έχουμε τα υδροελεκτρικά έργα. Δεν γίνονται όπως πρέπει ή κατασκευάζονται σε προστατευμένες περιοχές. Θα πρέπει η κυβέρνηση να υποβάλει ένα νέο πρόγραμμα δράσης που να αφορά και να καλύπτει και την ενέργεια. Αυτά θέλω να σας τονίσω, αλλά εν γέννη, μπράβο στον εισηγητή. Πολύ καλή συνεργασία. Ο επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην πρόταση ψηφίσματος για την ε, πρόοδο της Αλβανίας υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια σημεία, κάποιες ε, περιπτώσεις όπου αναφέρεται ένδειξη προόδου. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες αν μη τι άλλο αποδεικνύουν ότι η χώρα δεν δείχνει να ενδιαφέρεται και ιδιαίτερα στο να ανταποκριθεί στις απαιτήσει που έχει βάσει των ε, κανόνων και των υποχρεώσεων της συνθήκης Κοπενχάγης. Αυτές είναι πρώτα απ' όλα ο επεκτατισμός που φαίνεται από την υιοθέτηση της ιδέας Μεγάλης Αλβανίας μια κατάσταση η οποία στρέφεται κατά των συμφερόντων και των εδαφών υπάρχουν εδαφικές βλέψεις κατά των γειτονικών χωρών της Σερβίας, της Φύρομ, της Βουλγαρίας και της Ελλάδος. Αυτό παραβιάζει και την αρχή της καλής γειτονίας που υποχρεούται να επιδεικνύει η Αλβανία. Άλλη μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Αιγυπτίων, των Ρωμά αλλά και της ελληνικής μειονότητας του Βορείου Υπήρου που αριθμεί 300 περίπου χιλιάδες και κατοικεί στο νότιο τμήμα της χώρας. Εκεί παραβιάζονται ευθέω και τα θρησκευτικά δικαιώματα και τα πολιτικά, καθώς επίσης και τα δικαιώματα στην μόρφωση. Με την ανοχή του αλβανικού κράτους γκρεμίζονται ορθόδοξοι ναοί και υπάρχει μάλιστα η περίπτωση κατά την οποία ένας Έλληνας Αλβανός υπήκος ο οποίος έκτισε και πάλι ένα τέτοιο ναό να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της συλλήψεως και της φυλακίσεως. Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια να μην διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε μειωνοτικά σχολεία. Και επίσης καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ούτω ώστε πολιτικά να μην υπάρχει ελεύθερη δραστηριότητα των μειωνοτικών κομμάτων. Τέλος, υπάρχει αύξηση του Ισλαμιστικού εξτρεμισμού στη χώρα και έχει αυξηθεί ο αριθμός των ξένων μαχητών που αγωνίζονται κατά της Δύσεως και υπέρ του, του Άισις. Thank you very Σας ευχαριστούμε κύριε Επιτήδια. Το λόγο τώρα έχει η συνάδελφος Τάνια Φαγιών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ τον γιατί για την πολύ καλή και ισορροπημένη έκθεση. Τα πράγματα στην Αλβανία μπορούμε να τα δούμε υποθετικό πρίσμα σε ό,τι αφορά τις βασικές προτεραιότητες και θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημεία. Ένα τομέα ιδιαίτερος όπου θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια στη μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος. Το καλωσορίζω ως προτεραιότητα της κυβέρνησης και πόσο μάλλον που το αναγνωρίζει και η κοινωνία ως βασικό στοιχείο και θα πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση. Θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Υποστηρίζω επίσης και τις προσπάθειες του εισηγητή και άλλων συνοδέλφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την κατεύθυνση αυτή. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία, θα ήθελα να τονίσω την σημασία της διαδικασίας του Βερολίνου που αναφέρθηκε. σε ό,τι αφορά την ενέργεια, την νεολαία. Πολύ θετική αυτή η ατζέντα για την νεολαία και για την υπόλοιπη κοινωνία στην Αλβανία. Γιατί αν χάσει την ελπίδα της η νεολαία, χάνει το μέλλον τους οι χώρες και θα πρέπει να σταματήσει αυτό το brain drain, η διαφυγή εγκεφάλων στην περιοχή και μεταξύ της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αναφέρθηκε ότι αυτό αποτελεί μια μόνιμη οικονομική και πολιτική πίεση στη, στα μέσα ενημέρωσης που οδηγεί σε αυτολογοκρισία. Θα πρέπει να υπάρχει ένα υγιές περιβάλλον λοιπόν το οποίο θα δημιουργηθεί από την κυβέρνηση για τα μέσα ενημέρωσης. Ευχαριστώ πολύ Τάνια. Το λόγο τώρα έχει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γκέρακ Τσίγκερ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε έκθεση για την Αλβανία το 2015. Αποτίμησε τη σταθερή πρόοδο στον αφορά τι προτεραιότητε μεταρρυθμίσεων. Εκκρεμούν όμω μεταρρυθμίσει που πρέπει να γίνουν και θα πρέπει να γίνουν προσπάθειε που θα πείθουν από την Αλβανία. Αυτό αφορά κυρίω τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματο, κάτι που αναφέρθηκε επανειλημμένα σήμερα. Διεξοδική μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα αναμένεται να υιοθετηθεί του επόμενου μήνε και θα συμπεριλαμβάνει πλήρη έλεγχο του ποιοι διορίζονται ως εισαγγελείς και δικαστές θα είναι σαφές μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τότε η Αλβανία θα έχει καταβάλει αξιόπιστες προσπάθειες και η Αλβανία είναι έτοιμη να κινηθεί προς την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Όμως όλοι οι άλλοι τομείς των πέντε προτεραιοτήτων θα πρέπει και να συνεχιστούν. κατά Καταπολέμηση διαφθοράς, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, οι προσπάθειες θα πρέπει να αυξηθούν και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και αυτά θα πρέπει να ε, καλυφθούν. Και άλλες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν που δεν πρέπει να λησμονηθούν. Μερικές από αυτές αναφέρθηκαν εδώ. Ένα είναι η εφαρμογή ε, της, του νόμου περί αποποινικοποίησης που θετήθηκε το Δεκέμβριο αλλά η εφαρμογή θα πρέπει να ξεκινήσει σύντομα και αυτό θα δώσει άλλο ένα μήνυμα ε, ότι θέλει να προωθήσει τον επαγγελματισμό ε, στον επαγγελματικό τομέα Αλβανία και δεύτερον αυτό που αναφέρθηκε, δηλαδή οι συστάσεις του ελέγχου της εκλογικής διαδικασίας και ότι πρέπει να γίνουν εκλογικές μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Οι επόμενες εκλογές γίνονται σύντομα, τον Ιούνιο του 2017, οπότε θα πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος πολύ πριν ε, ξεκινήσουν οι εκλογές. Πολιτικοποίηση της διοίκησης του εκλογικού συστήματος και η πρόθεση της ε, διαφάνειας είναι κάτι που χρήζουν, χρήζει ιδιαίτερη ε, προσοχής το σχέδιο ψηφίσματο του κ. Φλεκενστάιν καλύπτει σωστά τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει του επόμενου μήνε η Αλβανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ τι εξελίξει και προσβλέπει στην οθέτηση αυτού του ψηφίσματο, διότι παρέχει περαιτέρω κατευθύνσει όσον αφορά ε, τι συνομιλίε και επαφέ με την Αλβανία στο εγγύ μέλο. Τεχνικέ και πολιτικέ συζητήσει με του συνομιλητέ στην Αλβανία θα συντηρηθούν, θα εντατικοποιηθούν του επόμενου μήνε θέλω να πω ότι θα κάνουμε διάφορες, ε, ε, διάφορες αποτιμήσεις ομολόγων. Θα, γίνει, θα συνεδριάσει η Υποπιτροπή ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του επόμενου μήνε και η κυρία Μογκερίνη, η πάτη εκπρόσωπο, αρχέ Μαρτίου θα επισκεφτεί τη χώρα και τέλο Μαρτίου θα γίνει διάλογο υψηλού επίπεδου για την ενταξιακή διαδικασία υπό την Προεδρία του Επιτρόπου Χάν και μετά θα γίνει και η συνεδρίαση των έξι υπουργών των Δυτικών Βαλκανίων αρχές Μαρτίου στα, στα Τύρανα. Συνεχίζεται η προσπάθεια ώστε να παρακολουθούμε συνεπώς και συνεχώς τις εξελίξεις και εξαρτάται την Αλβανία βεβαίως να δώσει αποτελέσματα, να δώσει αποτελέσματα βιώσιμα, αξιόπιστα, να δείξει ότι η χώρα είναι έτοιμη να προχωρήσει στην ενταξιακή διαδικασία. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριε Φλέγκενστάιν, θέλετε να πείτε λίγα λόγια. Μόνο λίγα λόγια και γερμανιστή. Λοιπόν, θα πρέπει να δημιουργηθεί, ε, να έχουμε διάφορα σημεία όπως είναι το περιβάλλον και άλλα θέματα που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, εκεί που χρειάζονται προσπάθειες δηλαδή. Ε, θα κινηθούμε λοιπόν και θα προσπαθήσουμε μαζί με τους κοιόδης να τα καλύψουμε αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις μεταρρυθμίσεις κοινωνικές και του εργασιακού, των εργασιακών συνθήκων θα πρέπει να δούμε τελικά φως στο τέλος της σύραγγας. Αν θέλουν να αναπτύξουν τη χώρα τους οι πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες. Χρειάζεται μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, είναι σημαντικότατες αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Εάν τελικά προωθηθούν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να συνεργαστούν επ' αυτού, διότι είναι συνταγματικής φύσεως οι αλλαγές, τότε αν γίνουν αυτά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συστήσει προς το Συμβούλιο την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να αναφέρω απλώς ένα σημείο που αφορά αυτά που είπε και ο Έλληνας συναδελφός μας. Είδαμε λοιπόν εδαφικές μεταρρυθμίσεις και Υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά τους Έλληνες της Αλβανίας. Αλλά η χώρα αυτή έχει πραγματικά πολλά προβλήματα. Αλλά πρόβλημα της ελληνικής μειονίτας όπως ε, παρουσιάστηκε, κανένας από τους συναδέλφους δεν μου το απέδειξε ότι υπάρχει και δεν μου το παρουσίασε και η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία γκρεμίστηκε, ήταν ένα γαράζ. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε τέτοια θέματα, προκειμένου να πραγματικά να μπορούμε να δρούμε. Αλλά η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη αρνητική μεταχείριση, διακριτική μεταχείριση. Θα είναι καλές λοιπόν ελπίζω οι συζητήσεις και ελπίζω να τελικά να καταθέσουμε μια έκθεση η οποία θα συγκεντρώσει μια ευρία Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Φλέκενστάιν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις προσπάθειες που κάνατε για την προετοιμασία της έκθεσης. Η Αλβανία είναι στην οδό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφώς έχει ορίσει κάποια benchmarks πρωτού ανοίξουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει και συμφωνώ ότι ο πολιτισμικός διάλογος και οι αντιθέσεις μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση, όχι μόνο για την Αλβανία, αλλά για όλε τι χώρε, αποτελεί βασική προπόθεση για να προχωρήσουν μπροστά. Θα υποστηρίξουμε λοιπόν τι προσπάθειε τη Αλβανία και θα παρακολουθήσουμε όλε τι εργασίε για τον σχηματισμό των σχετικών ε, επιτροπών. Τώρα, για τι προθεσμίε. 25 Φεβρουαρίου τη τροπολογία προθεσμία. 21 Μαρτίου θα γίνει η δεύτερη εξετασία εδώ στην Επιτροπή. Ψηφοφορία στις 21 πάλι με την φιλοδοξία να μπει στην Ολομέλεια του Απριλίου. Και τώρα περνάμε λοιπόν στο 12 της ημερήσιας διάταξης έκθεσης προ του 2015 για την Βοσνία και την Ερζεγοβίνη. Μοναδική ευκαιρία αυτή για μας, γιατί θα συζητήσουμε το πρώτο σχέδιο της έκθεσης του συναδέλφου του Κρίστιαν Νταν Πρέντα σε ό,τι αφορά την επίσημη η υποβολή υποψηφιότητα για ένταξη, την οποία επέβαλε χθε ε, στη Βοσνία, η Βοσνία και Ριζεγοβίνη στην ε, Ολλανδική Προεδρία του Συμβουλίου. Πάρα πολύ σημαντικό το βήμα αυτό από πολιτική άποψη για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη και ειλικρινά συγχαίρω τον πρόεδρο της Προεδρίας, όλη την Προεδρία, τους Υπουργούς Εξωτερικών και το καθεξής, όλους όσοι εμπλέκονται στην σημαντική αυτή διαδικασία. Η Ολλανδική Προεδρία τώρα θα θέσει αυτό το θέμα δεόντως στην ατζέντα του Συμβουλίου και θα ζητηθεί από το Συμβούλιο να γνωματοτήσει. Ξέρουμε ότι θα είναι μακρύς ο δρόμος για τη Βοσνία Ζεγοβίνη, μια χώρα η οποία ήταν θύμα επιθέσεων και έχει υποφέρει τα μάλα υπό το καθεστώς Μιλόσεβιτς. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για να προσεγγίσει τις Βρυξέλλες και υποστηρίζουμε λοιπόν τη διαδικασία αυτή με όλη μας την καρδιά. Μεταξύ άλλων ε, βασικός Παράγοντα από πλευρά του Κοινοβουλίου ήταν ο εισηγητή μα στη διαδικασία αυτή. Γι' αυτό λοιπόν να του δώσω το λόγο για να μα παρουσιάσει το σχέδιο τη έκθεση υπό το πλαίσιο των νέων ε, συνθήκων. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για την έκθεση, αλλά μια και η έκθεση έχει ήδη συζητηθεί ουσιαστικά, παρόλο που μας ονομάζουν οι συγητές, δεν είναι έκθεση αυτή που καταρτίζουμε εγώ και ο κύριος Τάνοκ ε, το έχουμε θίξει αυτό, αλλά δεν έχει επιληθεί το ζήτημα αυτό. Είναι, είναι η δεύτερη χρονιά που καταρτίζουμε τέτοιε εκθέσεις, οι οποίες ονομάζονται εκθέσεις, αλλά δεν αναγνωρίζονται από πλευράς ε, τεχνικής ως εκθέσεις. Αυτά για να σας υπενθυμίσω τι γίνεται ακριβώς. Όπως είπε λοιπόν και ο πρόεδρος της Επιτροπής, χθες ήταν μια σημαντική ιστορική στιγμή, 15 Φεβρουαρίου 2016, για την Βοσνία Ερζεγοβίνη, γιατί ο πρόεδρος ο οποίος ασκεί καθήκοντα πρόεδρο της ε, χώρας, επίσημα υπέβαλε την υποψηφιότητα της χώρας. Και να σας πούμε ότι στην έκθεση της Επιτροπής για μία φορά υπάρχουν και θετικά σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή οδό που ακολουθεί η χώρα. Και υπάρχει ασφαλώς μία σχέση μεταξύ της θετικής νότας αυτής και του, της ε, ιστορικής στιγμής που ζούσαμε χθε. Και είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε και να διαπιστώνουμε τις ε, ε, Φιλοδοξίας της ευρωπαϊκής και της κυβέρνησης αλλά και των πολιτών. Είναι μεγάλη στιγμή λοιπόν για την Βοσνία, μια στιγμή αισιοδοξία και για όλα τα αυτικά Βαλκάνικα. Βαλκάνια. Μια θετική στιγμή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, γιατί αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμα ένας πόλος έλξης του ευρωπαϊκού μοντέλου. Μια στιγμή όπου αυτό αμφισβητείται σημαντικά από μεγάλους φορείς ε, και στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όντως λοιπόν υπάρχει ένας πόλος έλξης. Είναι πολύ θετικό αυτό. Αλλά ας μην εθελοτυφλούμε. Είναι μια πρώτη αφετηρία, μια πρώτη φάση αυτή η κατάφαση της υποψηφιότητας. Από το εδώ και πέρα θα πρέπει να οικοδομήσουμε από πλευράς των αρχών της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους θα περιμένουν το καθεστώς της υποψήφιας χώρας. Θα έπρεπε να είμαστε ρεαλιστές και να υποστηρίξουμε το έργο το οποίο ήδη έχει γίνει. Να ανοίξουμε επίσης νέους τομείς εργασίας για να προσεγγίσει την Ευρώπη η χώρα. να μην ε, ε, εστιαστούμε μόνο στην ημερομηνία. Θα πρέπει να δούμε και το έργο που θα πρέπει να γίνει. Για το έργο λοιπόν αυτό θα πρέπει να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένο που θα πρέπει να ανθρωποποιήσω την παραγραφό 2 της έκθεσης σε ό,τι αφορά τους όρους ε, θέσης υποψηφιότητας, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ότι το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνής Αρζεγοβίνης στις 26 Ιανουαρίου ενέκρινε ένα μηχανισμό συντονισμού για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και στι 9 Φεβρουαρίου πάλι το Συμβούλιο αυτό ε, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για ε, ένα σύμφωνο συνεργασίας και σύνδεσης. Ε, αυτά τα δύο λοιπόν έπρεπε να επιληθούν ζητήματα και χαιρετίζουμε το γεγονός ότι μας πήραν στα σοβαρά, πήραν στα σοβαρά αυτές τις συστάσεις γιατί αυτό το είχε θέσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, όρο για την αξιοπιστία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης πέρα από την ατζέντα για τις μεταρρυθμίσεις που είχε συμφωνηθεί τον Ιούλιο του 2015. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες. Έχουμε καταρχάς το έργο του συντονισμού. Ο μηχανισμός συντονισμού θα πρέπει να προσαρμοστεί το στομότερο δυνατόν και αυτό αποτελεί σημείο κλειδί για την υποψηφιότητα της Βοσνίας Ερσεγοβίνης. και σε ό,τι αφορά άλλα ζητήματα. Οι διαπραγματεύσεις οι οποίες ε, συνεχίζονται σήμερα στο Σαράγεβο για τη Συμφωνία Σύνδεσης ελπίζουμε να σημειώσουν πρόοδο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 2013, είναι πάρα πολύ σημαντική για να επιτρέψει στη Βοσνία Ζεγοβίνη να προχωρήσει στις ε, μεταρρυθμίσεις ε, και σήμερα, μιας και είχαμε τόσο πολλά ζητήματα να συζητήσουμε, δεν θα ήθελα να επισέλθω σε υπερβολικές λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά το σχέδιο κειμένου, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια ζητήματα που μου φαίνονται πολύ σημαντικά η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνεται στην ατζέντα των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να συνεχιστεί για να βελτιωθούν οι κοινωνικονομικέ συνθήκε σε ό,τι αφορά του πολίτε τη χώρα. Η ανεργία, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, θα πρέπει να ληφθεί στα σοβαρά. Θα πρέπει, όπω πέρσι, να υπάρξει συνέχιση και των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στη Βοσνία Ζεγοβίνη προκειμένου να είναι δημοκρατικό κράτο, εύρυθμα λειτουργών. Η διαφθορά εξακολουθεί να είναι σε μεγάλα επίπεδα και μας ανησυχεί ιδιαίτερα και θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσει η καταπολέμηση της μάστιγας αυτής. Με τη βοήθεια των πολιτικών κομμάτων. Αν τα πολιτικά κόμματα δεν ε, σπρώξουν προς την κατεύθυνση αυτή, κανείς δεν πρόκειται να συνεχίσει τον αγώνα κατά της διαφθορά. Αν διστάσουν λοιπόν και κολυσιεργήσουν τα κόμματα αυτά, δεν θα ε, ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών. Οι πολίτες επίσης ζητούν μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, να μην υπάρχει πολιτική διάσταση σε ό,τι αφορά την απονομή της δικαιοσύνης, σε καταπολέμηση επίσης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Θα πρέπει να γίνει με πιο συντονισμένο τρόπο. Υπάρχουν ανησυχίε σε ό,τι αφορά την παρουσία των πυρήνων τρομοκρατίας στην χώρα. Επίσης, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνει υποχώρηση και η παναχώρηση σε θέματα ελευθερία τύπου. Και εκεί θα πρέπει λοιπόν να γίνουν σημαντικέ προσπάθειε γιατί τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση ε, αποτελούν τη ράχο κοκαλιά μια δημοκρατική κοινωνία. Και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για τη χρηματοδότηση των δημοσίων μέσων ενημέρωσης. Συναντηθήκαμε δε και με τους υπεύθυνους ε, διαχείρισης των δημοσίων αυτών υπηρεσιών και ακούσαμε αναλύσεις πολύ σοβαρές και για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την έκθεσή μου και αναμένω και τα σχόλια των σκιωδών και είμαι στη διάθεσή σας και ελπίζω να συνεργαστούμε όπως και πέρσι καλά προκειμένου και η τελική έκθεση να βρει την υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά, κυρία Πρέντα. Δίνω τον λόγο στον φίλο Φεσκάν που είναι ο σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον συνάδελφο τον Κρίστιαν Πρέντα. Είναι ισορροπημένη η έκθεση πρόοδου για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Χτες γιορτάσαμε την επίσημη αίτηση της χώρας που υπέβαλε για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωατλαντική ολοκλήρωση είναι η καλύτερη ελπίδα για σταθερή και ευημερούσα Βοσνία. Μακρύ το ταξίδι που θα ακολουθήσει η χώρα. Όμως σημαντικό το ταξίδι. Η πρόοδος της Βοσνίας είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι θέλουμε σταθερότητα και ευημερία στη γειτονιά μας. Χαίρομαι που η Βοσνία τώρα έχει μηχανισμό συντονιστικό που βρίσκει τρόπους για διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά μαντάτα αυτά. Πρέπει να δούμε όμως πώς λειτουργεί στην πράξη ο μηχανισμός αυτός. Ανησυχώ για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε ο μηχανισμός. Δεν υπήρξε διαβούλευση με μέλη αντιπολίτευσης, ούτε με την κοινωνία των πολιτών, ούτε με τους πολίτες. Φαίνεται ότι ο μηχανισμός επίσης δίνει μεγάλες δυνατότητες λήψης αποφάσεων στα καντόνια στους διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που μπορεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις και να τις κάνει περίπλοκες. Και αποδυναμώνονται τα διάφοροι θεσμοί του κράτους. Και επίσης η νομολογία του Δικαστηρίου της Βοσνίας ε, και του Εθνικού Εισαγγελέα ανησυχεί. Στα πλαίσια του διαθρωμένου διαλόγου η δικαιοσύνη πρέπει να εργαστούμε σκληρά για πιο αποπολιτικοποίηση των θεσμών εάν δεν γίνει σεβαστό το κάτω δικαίου και δεν υπάρχει λογοδοσία στο δικαστικό τομέα, θα αποτύχουν όλες οι άλλες προσπάθειες. Συμφωνώ απόλυτα με τους ηγητές ότι τα κοινωνικονομικά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να έχει προτεραιότητα αυτό. Θα πρέπει να είναι υπόλογη η κυβέρνηση να αφορά τι μεταρρυθμίσει δημόσια Θα υποστηρίξουμε πρωτοβουλίε να δημιουργηθεί ένα κλίμα θετικό για τι επιχειρήσει και για την ανταγωνιστικότητα στη Βοσνία. Θα πρέπει να πιέσουμε για κοινωνική ευημερία, μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και του συνταξιδοτικού. Αυτό χρειάζονται και θέλουν οι Βόσνοι. Θα πετύχουμε μόνο όταν οι πολίτες αρχίζουν να ωφελούνται άμεσα από τις προσπάθειες εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Και τότε αρχίζει να διαμορφώνεται μια ευρωπαϊκή Βοσνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα να δώσω το λόγο, εφόσον δεν βλέπω συναδέλφους του ECR, στον κύριο Ράντεσ της ε, Άλντε. Έχετε το λόγο, συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Πρέντα, πληρέστατη έκθεσή του. Και τον ευχαριστώ για όλα όσα κάνει συνήθως πέρα από τις υποχρεώσεις που έχει ως εισηγητής. Προσπάθειες που κάνει να προωθήσει την ευρωπαϊκή πορεία της Βοσνίας Ζεγοβίνης. Πριν υποβάλει το αίτημά τη για να γίνει μέλος η Βοσνία Ζεγοβίνη, οθέτησε στη σημαντικότατα έγγραφα. Το πρώτο είναι ο συντονιστικός μηχανισμός και το άλλο είναι το σχέδιο διαπραγματεύσεων. Ή μάλλον το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την προσαρμογή της σχετικής συμφωνίας. Πρόσφατα πριν υιοθετηθεί το σχέδιο μεταρρυθμίσεων για το 2015 μέχρι το 2018, υιοθετήθηκε ένα ενδιάμεσο σχέδιο δράσης για να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις. Φαντάζομαι ότι το πλούστερο έγγραφο και το ευκολότερο θα ήταν η προσαρμογή της σχετικής συμφωνίας που έχει συναυθεί, διότι φαντάζομαι ότι μέχρι τώρα αυτό δεν ήταν κάτι υποφελές για την κυβέρνηση και τώρα έγινε το τεράστιο βήμα πρόοδου και είναι σημαντικό τα διάφορα θέματα να καλυφθούν. Όμω η λειτουργία του συντονιστικού μηχανισμού με τις ε, περιπλοκές που ανέφερε ο κύριος Καν και η εφαρμογή του μεταθυσμικού σχεδίου θα είναι δυσχερέστατα τα πολιτικά έργα προς επιτέλεση. Να αναφέρω μια διάσταση όσον αφορά το μεταρρυθμιστικό σχέδιο για να σας δείξω πόσο τεράστιο πρόβλημα έχει να αντιμετωπίσει η Βοσνία Εζεγοβίνη. Είναι η εξυγίανση δημοσιονομική του κράτους και ε, να μειωθεί η γραφειοκρατία η κρατική. Η μείωση των δημοσίων δαπανών που όπως αναφέρεται στο σχέδιο συνεπάγεται μεταρρύθμιση Άρα, μείωση ίσως των συντάξεων της ε, περίθαλψης της υγειονομικής και όλα αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να περάσουν χωρίς πολύ σοβαρές προσπάθειες ή αντιμετώπιση δυσκολιών για να διατηρηθεί ταυτόχρονα και η κοινωνική συνοχή στην όλη προσπάθεια. Η Βοσνία Ζεγοβίνη αντιμετωπίζει περιπλοκότατο, δυσχερέστατο δρόμο. Χτες έκανε τεράστιο βήμα προόδου, αλλά πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί ε, στις ανάγκες αυτές η ε, Βοσνία Ζεγοβίνη. Θα προσπαθήσουμε μέσω τροπολογιών εμείς να συμβάλλουμε στην όλη πίωση ε, της προσπαθίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέσεριτς και μετά Κροατία και Σλοβενία θα πάνε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδης εισηγητής για αυτό το θέμα, αλλά συνάδελφος ο Ίγκορ Σόλτες Έφυγε. Έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Η Ζουγκάντα ως παρατηρητής εκλογών χαιρετίσματα στέλνει στον συγγητή και θέλει να διαβάσω ότι είναι πολύ ικανοποιημένο με την έκθεση. Είναι πάρα πολύ περιεκτική και σύντομη, όμω πολύ ουσιαστική στο περιεχόμενό τη. Θα ήθελα να προβώ σε δύο γενικά πολιτικά σχόλια και μετά κάποιε λεπτομέρειε να αναφέρω. Νομίζω ότι η υποβολή του αιτήματο ένταξη από πλευρά κυβερνήσεω τη Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι κάτι ευπρόσδεκτο. Εμεί, σαν Ευρωκοινοβούλιο, θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη τώρα να εξετάσουν με ενεργό τρόπο το αίτημα αυτό τη ένταξη τη ε, Βοσνία Ερζεγοβίνη να στείλουν το ερωτηματολόγιο του το ταχύτερο δυνατόν, ώστε η όλη διαδικασία να ξεκινήσει πραγματικά. Ταυτοχρόνως όμως είναι σαφές ότι η υποβολή της αιτήσεως δεν σημαίνει ότι πληρούνται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις και ότι έχουν γίνει ε, και έχουν υλοποιηθεί οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Είναι μακρύς ο δρόμος για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Αναφέρθηκε η συνταγματική μεταρρύθμιση και η νομική μεταρρύθμιση και στη συνταγματική μεταρρύθμιση έχουμε ακαθόδες θέμα δηλαδή ε, ότι το παρόν σύνταγμα εμποδίζει τις πολιτικές ε, εξελίξεις στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Αν η Βοσνία θέλει να προχωρήσει και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα που απομακρύνεται από την εκδοχή του Dayton και να δώσει ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες και όχι μόνο σε εθνοτικές ομάδες. Αυτό είναι άκρος ευαίσθητο θέμα για τη Βοσνία Ζεγοβίνη και πρέπει να εξεταστεί προσεκτικότατα. Δεύτερον, εντός του, της μεταρρυθμίσης του δικαστικού τομέα με κάτι. Τι γίνεται με τα εγκλήματα πολέμου και χρήση εναλλακτικών μεθόδων για τη μεταβατική δικαιοσύνη. Κάτι που θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Τίποτα δεν εφαρμόζεται από τις συστάσεις που έγιναν από τις αρμόδιες φορείς του ΟΗΕ για τη δικαιοσύνη στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Και κάτι άλλο. Ο νόμος για την νομική αρρωγή ε, ήταν στο, στην ατζέντα για το εθρομένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει την προτεραιότητα. Πρέπει να δοθεί η προτεραιότητα. Είναι ένα τμήμα σημαντικό της μεταρρύθμισης του δικαστικού τομέα. Πρόσβαση στην νομική αρρωγή, στις νομικές υπηρεσίες είναι ένα βασικό στοιχείο στο κράτος δικαίου. Τέλος, να επαναλάβω ότι η έκθεση είναι σύντομη αλλά περιεκτική, περιέχει πολλή ουσία. Ε, και πιστεύω ότι η συνάδελφος ε, θα έχει άριστη συνεργασία με τον εισηγητή. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, αγαπητέ συνάδελφοι. Message. Και τώρα, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κασούτσα, που είναι ε, η ε, αντιπρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας για τη σχέση με τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον φίλο Κριστιαν Πρέντα, διότι είναι εξαιρετική η δουλειά του και αυτό το κείμενο, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει τώρα με τη καινούργια συγκυρία, πώς θα, πώς θα αλλά δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε την χθεσινή ημέρα που ήταν ιστορική για την Βοσνία Ερζεγοβίνη, ε, πάρα πολύ σημαντική για την ε, ευρωπαϊκή της ε, και ατλαντική της πορεία, διότι απετέλεσε καρπό αυτής της γενιαίας προσπάθειας από την Προεδρία, από όλες τις πολιτικές πτέρυγες σε σχέση και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να με τα καλύτερα στη χώρα αυτή. Αλλά όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας στην Ανατολική Ευρώπη, είναι αυτό μια υπόθεση πάρα πολύ σημαντική, ούτω ώστε να δοθεί συνέχεια σε αυτή την ευρωπαϊκή διαδρομή και γι' αυτό και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόκειται να δώσει τη σχετική εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να γνωμοθετήσει, να ξεκινήσει η διαδικασία τη πρόσβαση και η Βοσνία να γίνει υποψηφία χώρα αφού θα λάβει το πράσινο φως που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χθε ε, ο κ. Χάνη και οι συνάδελφοι αλλά και η κυρία Μογκερίνη συνεφώνησαν ότι πρόκειται για μια σοβαρή υποψηφιότητα. Και ε, σήμερα στο Σαράγεβο συνεχίστηκαν οι δύο πραγματεύσεις, ελήφθησαν πολλά προβλήματα ε, επικαιροποιήσαμε την προηγουμένη συμφωνία, συγκροτήσαμε μηχανισμούς συντονισμού που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, νομίζω ότι ορίμεσαν τα πράγματα για τη χώρα αυτή. Οπότε, τώρα την ε, σκητάλη ε, έχει η ηγεσία της χώρας, οι διάφοροι θεσμοί. Είναι μονόδρομος η ένταξη για τη χώρα αυτή, οπότε και θεωρώ ότι ε, θα δουλέψει το μοντέλο το ομοσπονδιακό και η αποκέντρωση στη χώρα θα αποδώσουν. Ε, επίσης το Κοινοβούλιο αλλά και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θεματολογιό τους θα κρατήσουν την ένταξη της χώρας υψηλά. Όλοι θα συμβάλλουν για αυτή την πορεία. Και βέβαια είναι πρόβλημα η τρομοκρατία. Βέβαια εκεί υπάρχει έφορο έδαφος για τους τρομοκράτες. Αυτό δεν το ξεχνάμε υπάρχουν και προβλήματα με τα μέσα ενημέρωση σε όλη την περιοχή αυτή της Ευρώπης, ε, κύριε Πρέντα. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη χρηματοδότηση των κρατικών ΜΜΕ. Υπάρχει θεματολόγιο μεταρρύθμισης, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούν στα σοβαρά. Πάντως, βλέπουμε θετικά τα πράγματα, θα πρέπει να δουλεύει σκληρά η χώρα. Μα κοιτάξτε και η Κροατία πριν από λίγα χρόνια πήρε το πράσινο φως από τότε που έγινε και η υπογραφή των σχετικών εγγράφων. Κράτησε σχετική δρομή 8 χρόνια, μπορεί να μην κρατήσει τόσο για τη Βοσνία, αλλά θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι είναι σοβαρή δουλειά που κάνανε και άρα θα πρέπει να επιληθούν όλα τα πολιτικά θέματα τα οποία εκκρεμούν και να βελτιωθεί και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Αλλιώς, αλλιώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα την χώρα. Άρα, εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε αυτή τη χώρα, να υποστηρίζουμε τις αλλαγές που γίνονται εμείς όλοι στην Επιτροπή μας. Ο κύριος Πίτσουλα τώρα, λέει ο πρόεδρος, έχετε τον λόγο, Πίτσουλα. Θα πρέπει να συγχαρούμε τον κύριο Πρέντα. Είναι εξαιρετική η έκθεσή του. για την ε, πρόοδο την τελευταία χρονιά της χώρας. Ήταν εξαιρετική αυτή η χρονιά, ξεχωριστή από πλευρές απόψεις και βεβαίως υπάρχει μια έγγραφη δέσμευση όλων των πολιτικών ηγετών της χώρας όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Έτσι προβλέπει και η Συμφωνία Σύνθεσης. Οπότε η, πρόεδρος, η πρόοδος της χώρας ξεκίνησε πέρσι, τότε που υπέβαλαν την αίτηση ένταξης, να επομένως απόδειξη του πόσο χρειάζεται να αλλάξουν τα πράγματα από τότε που ξεκίνησε το κύκλο ζήτηση αυτή τη χώρα, από τη συμφωνία του Ντέιτον μέχρι τη συμφωνία των Βρυξελών και είδαμε τώρα πώς βελτιώνονται οι επιδόσεις τους. Δεν θα πρέπει να αμελούμε το τι χρειάζεται να γίνει για την ένταξη. Πρώτα πρώτα, αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε υλοποίηση αυτού του μηχανισμού του συντονισμού. Να συνεχιστεί το θεματολόγιο της ε, μεταρρύθμισης θα πρέπει να υλοποιηθεί η Συμφωνία Σύνδεσης ε, επίσης πρέπει να γίνουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις και θα πρέπει να γίνει πιο λειτουργικό το πολιτικό σύστημα χρειάζεται και διοικητική μεταρρύθμιση δεν έχει γίνει θα πρέπει να υλοποιηθεί ο ομοσπονδιακός χαρακτήρας και η επικουρικότητα. Βέβαια, δεν είναι όλοι στη χώρα το ίδιο ενθουσιώδες. Δεν είναι όλοι το ίδιο όριμοι για μεταρρυθμίσεις. Υπήρχε πρόβλημα στο Κοινοβούλιο. η Εθνική Συνένεση δεν ήταν δεδομένη. Όμως υπάρχουν διάφοροι παράγοντες μέσα στη χώρα και έξω από αυτήν, ώστε να βοηθήσουν ε, στην μεγάλη αλλαγή. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν την ύφη οι πολίτες. Έχουμε 62% ανεργία στους νέους και πάρα πολλούς μακρόχρονα ανέργους. Να, πώς φαίνεται το πρόβλημα της οικονομίας. Επίσης, υπάρχουν κάποιες εθνοτικές ομάδες που δεν έχουν ίδια δικαιώματα όπως όλοι οι υπόλοιποι. Πάντως, υπάρχει σίγουρα κάποια πρόοδος. Μαριάννα Πετήρ, Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει κυρία Πετήρ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια στον κύριο Πρέντα πάρα πολύ λεπτομερής και ισορροπημένη έκθεση. Να συγχωρούμε επίσης και τη Βοσνία Σεγοβίνη, η οποία ζήτησε υπέβαλε υποψηφιότητα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε στο μέλλον της Βοσνίας Ερσεγοβίνης και πιστεύουμε ότι η Βοσνία Ερσεγοβίνη έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα προς ένα μέλλον όπου και οι τρεις λαοί θα ε, έχουν τις ίδιες αξίες, τις ίδιες ευκαιρίες. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει ακόμα σήμερα. Σήμερα οι Κροάτες αποτελούν ε, έναν από τους λαούς που συναποτελούν την Εγγλική Ριζεκοβίνη μόνο στα χαρτιά. Τα ανθρώπινα δικαιώματά τους παραβιάζονται και δυστυχώς έχουν εκλείψει πλήρως από κάποια τμήματα της Βοσνίας Ριζεκοβίνης. Και είναι η ιδιαίτερη σχέση των μέσων ενημέρωσης ε, της χώρας με την κρατική κοινότητα. Είναι σημαντικό λοιπόν να σας προειδοποιήσω να αλλάξει αυτή η τρέχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά και την κρατική γλώσσα, γιατί η κρατική γλώσσα δεν είναι επαρκώς παρούσα στα μέσα ενημέρωσης. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω το εξής. Δυστυχώς δεν υπήρξαν ε, βελτιώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος και της ε, διασυνοριακής ρήπανσης και το τι συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον. Και έτσι ο κόσμος υποφέρει ακόμα από τα δηληστήρια που λειτουργούν κοντά στα σύνορα. Και στα σύνορα με την Κροατία πολλά από τα έργα που διεξαγάγονται θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον της Κροατίας. Αυτό κατά παραβίαση όλων των ε, συνθήκων τις οποίες έχει που γράψει η Βασνία Ζεχοβίνη. Θα ήθελα λοιπόν ο εισηγητής να δώσει ιδιαίτερη σημασία και σε αυτή τη σημαντική ψυχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαριάννα. Και τώρα να περάσουμε στη Σλοβενία. Τάνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για την ισορροπημένη έκθεση και ήδη χθε ανέφερα ότι έξι χρόνια και πλέον μετά από την κατάργηση του καθεστώτος της, ε, των θεωρήσεων, η Βοστία Ζεγοβίνη έκανε ένα σημαντικό βήμα για νέες ευκαιρίες για τη χώρα. Αυτό ασφαλώς εξαρτάται και από τις μεταρρυθμίσεις ε, που με τη σειρά τους εξαρτώνται από τους πολιτικούς της χώρας. Ε, ελπίζω η χθεσινή ημέρα η οποία θα περάσει στην ιστορία, να δώσει ένα νέο κίνητρο για το μέλλον. Εύχομαι λοιπόν κάθε επιμέλεια και κάθε κουράγιο προς ε, την χώρα. Αυτό θα καθορίσει άλλωστε και την ταχύτητα της εισχώρησης στην Ένωση. Να υπογραμμίσω όμως το θέμα των μέσων ενημέρωσης, το θέμα ιδιαίτερος της ύπαρξης ε, του Εθνικού Σταθμού DHRT. Ο, η μοναδική εταιρεία μέσων, μέσων ενημέρωσης, η οποία τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ήταν το τελευταίος δημόσιος σταθμός. Αν καταργηθεί και αυτός, θα μιλάμε για τρία κράτη σε ένα. Πλέον. Και θα υπονομευτεί η ύπαρξη της χώρας. Να ρωτήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ακριβώς συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάνια. Ο κύριος Πέτερλε τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μολτσουμέσκ, κύριε Πρέντα. Καλώς ορίζω την επιθυμία του εισηγητή να καταστούν πραγματικές εκθέσεις ή εκθέσεις πρόοδου. Και χαίρομαι που αυτή η καλή έκθεση πραγματικά αναφέρει μία πρόοδο. Μία αλλαγή στην στάση, αν θέλετε, από πλευρά τη βοσνιας Ριζεγοβίνη σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλώ ορίζω στο πλαίσιο αυτό και την καλή θέληση μετά τη χθεσινή ημέρα σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητα, το σχεδίο δράσης, το, το μηχανισμό συντονισμού στα διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Αυτό πιστεύω αποτελεί μία βάση για έναν κοινό παρανομαστή για την προσέγγιση της Βοσνής Ρεζεγοβίνης στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα τα υπόλοιπα τα είπαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Πλένκοβιτς. Το λόγο έχει ο κύριος Σίγκλερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως θα συνεχίσετε στα σλοβενικά ή στα κροάτικα. Θα ήταν ε, ενδιαφέρον. I could do it in Polish, but... Θα μπορούσα να το κάνω πολωνικά, αλλά σε άλλες γλώσσες δεν μπορώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την επίκαιρη αυτή συζήτηση μετά την ιστορική υποβολή ετήσους ε, ένταξης. Ε, λοιπόν, έτσι εκφράζονται οι προσδοκίες του λαού της Βοσνίας Αζεγοβίνης να κινηθούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνει ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι ικανό να μπορέσει να πετύχει τα αποτελέσματα από τη στιγμή που όλοι οι ηγέτες και ό, σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα μπορούν να συνεργαστούν προς τον κοινό στόχο. Βεβαίως αυτό σημαίνει αντιστρόφως ότι αν αυτοί οι ηγέτες σε διάφορα επίπεδα δεν συνεργαστούν, τότε το σύστημα θα λειτουργήσει. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάποια επιτύγματα του τελευταίου δεκαμήνου, κάποια από αυτά αναφέρθηκαν εδώ. Ε, τέθη η συμφωνία σε εφαρμογή πέρσι, μεγάλο βήμα μετά από 7 χρόνια προσωρινή συμφωνία. Μετά έγινε το πρώτο συμβούλιο και η πρώτη επιτροπή συνεδρίαση στο τέλος του 2015 και μετά τον Ιούλιο πέρσι είχαμε την έγκριση του θεματολογίου, της μεταρρύθμισης, αρχή της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και αυτό που προαναφέρθηκε εδώ είναι ότι σήμερα δόθηκε νέα ε, διαπραγματευτική εντολή για τη συνέχιση της διαδικασίας αλλά θα αναφερθώ στα ήδη υποθέντα ότι στην επανάληψη τώρα των συνομιλιών όσον αφορά τις αναγκαίες προσαρμογές βρίσκουμε απλώς την αφετηρία και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέρμα της διαδρομής και τέλος η οθέτηση του μηχανισμού του συντονιστικού είναι κάτι που αφορά τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, να δούμε τι γίνεται στην πραγματικότητα, θα γίνει η δοκιμή και ήδη αμφισβητείται ο μηχανισμός από τη Ρεπούμπλικα Σέρτσκα και θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα στην πράξη πριν γίνει η αξιολόγηση η ηγεσία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την ορμή που έχει δημιουργηθεί και να εργάζεται σκληρά η πρόοδος και η υλοποίηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων είναι και κάτι που ανταποκρίνει στις προσδοκίες ε, του λαού και είναι προϋπόθεση για το επόμενο βήμα, άρα το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί όσον αφορά την ε, υποψηφιότητα αυτή. Αυτό είναι σημαντικό βήμα που θα λάβει η χώρα από τη στιγμή που θα έχει σημειωθεί ε, επαρκής προόδος στον φορά Και έτσι θα κάνουμε τα δέοντα και θα λειτουργήσει ο διευθυντικός μηχανισμός. Είναι σημαντικό λοιπόν οι μεταρρυθμίσεις να πραγματοποιηθούν σε στενή συνεργασία με τους διεθνείς χρηματοστατικούς μηχανισμούς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί μαζί με αυτούς τους φορείς εκ του σύνεγγυς τις μεταρρυθμίσεις και θα στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις στο βαθμό του δυνατού. Τώρα όσον αφορά την ε, έκθεση, το ψήφισμα μάλλον, του κυρίου Πρέντα, τον ευχαριστούμε πολύ. Θεωρούμε ότι τρίζει άριστα τα προβλήματα, ισορροπημένη έκθεση και ταυτίζεται και με τα πορίσματα της εκθέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει όλος ιδιαίτερος την υποστήριξη που παρέχει το ψήφισμα για το επόμενο βήμα του μονοπατιού της ένταξης της χώρας κυρίως όσον αφορά την ανάγκη η χώρα να συνεχίσει με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων μέσω των τριών πυλώνων κοινωνικονομικό πυλώνας, κράτο δικαίου και δημόσια διοίκηση αυτήν τη πυλώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίλερ. Κρίστιαν, θέλετε να πείτε κάτι. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους. Για τις, ε, τα σχόλια τους και τις δράσεις τους. Και προφανώς ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη η ανταλλαγή απόψεων, γιατί μπορώ έτσι να προβλέψω κάποιες από τις τροπολογίες που θα κατατεθούν. Αυτό είναι θετικό. Θα πρέπει να διευκρινίσω ότι και εγώ ο ίδιος έχω τροπολογίες να καταθέσω, δεν το έκανα δεδομένων και των περιορισμών σε ό,τι αφορά την έκταση του κειμένου. Στη συνέχεια θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος στην Βοσνία Ερσεγοβίνη. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε συμβιβασμού ε, πιο περίπλοκους από ό,τι μπορεί καν να φανταστεί κανεί εκ πρώτη όψεω. Και προφανώς ε, αυτό το παραδέχονται και οι και το παραδέχονται και οι φίλοι της ευρωπαϊκής προοπτικής ε, της Βοσνής Ερζεγοβίνης. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα, γιατί υπάρχουν κάπως περίεργες πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλία συγκεκριμένα που παρουσιάζονται ως δημοκρατικές για να μπλοκάρουν τη δημοκρατική πορεία. Τα δημοψηφίσματα, τα δημοψηφίσματα τα οποία προτείνονται από τους ε, ηγέτες της Ρεπουμπλικά Βυσέρευσκα για να μπλοκάρουν την ευρωπαϊκή πορεία, το δημοψήφισμα ε, για να μπλοκάρει την πορεία αυτή της χώρας δεν είναι κάτι που εφήβρε η Ρεπουμπλικά Σέψχα. Το είδαμε και στην Κρυμαία από τον ε, Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας και ο Ματιέντεφ το τόνισε ότι δεδομένου του δημοψηφίσματος ε, επιβεβαιώνεται το μέλλον της Κρυμαίας. Ε, ο ίδιος δρόμος ακολουθείται. Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν είναι εφεύρεση της ε, Ρεπουμπίξκα, Σέρψκα. Από αυτή λοιπόν την άποψη, η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να είναι πολύ πιο αμήλικτη. Γιατί πρόκειται για το μέλλον, το μέλλον ενός ευρωπαϊκού λαού. Αυτό διακυβεύεται. Άρα χρειάζεται θάρρος και τόλμη. Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε την πραγματικότητα η οποία πραγματικά είναι ξεκάθαρη. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους για τις απαντήσεις τους και για την αντίδρασή τους και χαίρομαι που δεν το βλέπετε σε ένα γραφικό θέμα το θέμα της, πολιτι... της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης αλλά ως ένα θέμα πολιτικά κρίσιμο. Ευχαριστώ. Κρίστιαν, λέει ο Πρόεδρος, πολύ καλή η συζήτηση και προσβλέπω στην κατάθεση τροπολογιών από πλευράς των συναδέλφων. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να κινηθεί γρήγορα και σταθερά η Βοσνία Ζεγοβίνη στην πορεία προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι πεπισμένος ότι η κατάσταση της υποψηφιότητας χτες θέτει απαραίτητα τον ρυθμό που θα ακολουθήσει η χώρα και θα είναι και το τελικό συμβατικό στοιχείο για τη χώρα, αν θέλετε, θα δώσει μια αποστομωτική απάντηση σε όλους τους αποσχιστές και θα επιτρέψει και στις τρεις κοινότητες και σε όλους όσους ε, ζουν στη Βοσνία Ζεγοβίνη να είναι ίση. Και όταν θα έρθει η στιγμή της δεγματικής μεταρρύθμισης να μετακινηθούν από τη Συμφωνία Dayton που ισχύει σήμερα. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν στη σημερινή συζήτηση και η κατάθεση για τροπολογιών είναι μέχρι 29 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. 21 Μαρτίου η ψηφοφορία, 22 Μαρτίου, 21 ε, Μαρτίου δεύτερη εξέταση, 22 η ψηφοφορία στον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Επόμενο θέμα, το 13 της σας διάταξης. Πολύ σημαντική έκθεση. Μία από τις εκθέσεις κλείδι για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, ένας πιο συνδεδεμένος και πολύ σύνθετος κόσμος. Η Σάντρα Καλνιέτα είναι η συγγητριά μας, έχει γίνει πριν από κάποιες εβδομάδες η πρώτη ανταλλαγή απόψεων όπως ε, όλοι σας εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο το οποίο είχε ήδη ολοκληρωθεί δεδομένων και των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο Και πριν η κυρία Μογκερίνη παρουσιάσει τον Ιούνιο τη νέα της έκθεση στο Συμβούλιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με σαφήνεια περιγράφονται όλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως παγκόσμιος παράγοντας στην ε, ανατολική και νότια γειτονιά μας. Ποιες θα είναι οι αρχές μας, οι αξίες μας, τα μέσα με τα οποία προτιθέμεθα να προσπιστούμε τις αρχές αυτές στην παγκόσμιο προσκήνιο για να ενισχύσουμε την εξωτερική μας δέσμευση. Και τώρα ασφαλώς θα δώσω το λόγο στην κυρία Καλνίατα για να μας πει τι γίνεται και σε ποια φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την έκθεση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφε, θα έχετε λάβει το σχέδιο κειμένο όσον αφορά ακριβώς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο και μετά όλες τις συνοήσεις, συμβιβασμούς και διαπραγματεύσεις καταλήγουμε σε ένα δυναμικό κείμενο το οποίο αντικατοπτρίζει τη θέση του Κοινοβουλίου για μια παγκόσμια σφαιρική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πάει στην Ολομέλεια τον Απρίλιο και ευχαριστώ τους συναδέλφους στην ε, Επιτροπή γιατί οι προτάσεις τους ήταν ε, πάρα πολύ αξιόλογες. Ίδιος, την κυρία Μισελόλιο Μαρή, την ευχαριστώ για τις αξιόλογες συμβολές της στο σχέδιο του κειμένου. Όλοι γνωρίζουμε ότι το να χαράξει κανείς μια παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική μας πολιτική είναι κάτι το δύσκολο αλλά πολύ χρήσιμο γιατί ε, ακόμα υπάρχει απόκληση στο τι θέλει κάθε μέλος και λέμε ότι καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η θέση να γίνει εταίρος στρατηγικός. Οπότε γι' αυτό ας εξετάσουμε τους εσωτερικούς φραγμούς. Και πρώτα-πρώτα έχω να σας πω ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση ούτως ώστε να ενεργήσουμε από κοινού ως Ένωση και να χρησιμοποιήσουμε όλες μας τις δυνατότητες, όλα τα εργαλεία που έχουμε ούτως ώστε να πετύχουμε τους στόχους της πολιτικής μας. Αλλά υπάρχει και το θέμα της ε, δαπάνης της πολιτικής μας. Δεν υπάρχει συνεργασία, δεν υπάρχουν συνέργειες όσον αφορά τις σχετικές ε, σχετικούς διαγωνισμούς και επίσης μεταξύ άλλων δεν υπάρχει αρκετή συνέπεια στις εξωτερικές και εξωτερικές πολιτικές. Όλοι γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα οποία επισημώνονται στην στρατηγική του 2003 ε, συνεχίζουν όλα αυτά να είναι επίκαιρα έχουμε όμως και νέες προκλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κυβερνοέγκλημα, ας πούμε, αλλά την μετανάστευση, την αλλαγή του κλίματος. Όλα τα τροτά σημεία και αδυναμίες μας. Υπάρχει αναφιωρητική τάση που θέλει να ανατρέψει τα πράγματα. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται με αυτές τις λεπτές δημογραφικές και όχι μόνο ισορροπίες. Επίσης, Πρέπει να σας πω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε για Ασία και Ειρηνικό έχουν αναθεωρήσει τις προτεραιότητές τους. Για ασφάλεια κυρίως. Επίσης, έχουμε τώρα αυτό το σχεδίο κειμένο, τα έχουμε πει με τους συναδέλφους και θα πρέπει να βρούμε απαντήσεις στο ποια είναι τα στρατηγικά μας συμφέροντα, ποιες οι προτεραιότητες της εξωτερικής ε, δράσης και τι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλεία και τι πόρους. Τι προσέγγιση να έχουμε για αυτή την εξωτερική δράση. Θέλω να συνδυάσω στο κείμενο την γεωγραφική προσέγγιση και την θεματική. Να θέσουμε κάποιες προτεραιότητες και στόχους. Τέλος, θεωρούμε ότι αυτές οι τρεις προτεραιότητες που υπάρχουν μπορούν να καλύψουν περισσότερους στόχους. Ποιες είναι οι προτεραιότητες. Πρώτα πρώτα. Άμυνα και προστασία αξιών χωρών και κοινωνιών. Και αυτό να καλύπτει όλη την Ευρώπη και τους γείτονες μας. Σημαίνει αυτό επίση ότι θα πρέπει κάπω να αναπτύξουμε κάποιε δυνάμει ευρωπαϊκέ που να δρούν συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ όσον αφορά την άμυνα τη υπηρεσία μα και να μπορούμε να έχουμε κάποιε επιχειρήσει ε, και επεμβάσει πέρα των συνόρων τη Ευρώπη, τώρα κάτι άλλο το οποίο προτείνω είναι να μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάποια σταθερότητα όσον αφορά την ε, ευρύτερη ε, περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ολένα και περισσότερη ε, συνεργασία επί τη βάση της ε, διεύρυνσης και επί της ε, διαχείρισης των κρίσεων, παρέμβαση και διαχείριση κρίσης, εξωτερική δράση και εσωτερική ασφάλεια. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την οικονομική συγκυρία, τι τα θέματα ταυτότητας, τα θέματα ασφάλειας. Κάτι άλλο το οποίο σας προτείνω είναι ότι θα πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται σε παγκοσμία κλίμακα, πώς θα έχουμε μια παγκόσμια διακυβέρνηση, εμπόριο, το οικονομικό σύστημα, την αλλαγή του κλίματος, ε, τον κυβερνό χώρο, αλλά επίσης να δούμε πώς γίνεται η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τι γίνεται με την λάθρομετανάστευση, τι γίνεται με τη μετεγκατάσταση των προσήγων και τι γίνεται σε σχέση με την Αφρική που έχουμε πολλά εργαλεία και αυτά ενσωματώνονται στις ε, συνθήκες αλλά, αλλά δεν έχει γίνει σωστή υλοποίηση των όσων προβλέπονται ή δεν τα έχουμε αξιοποιήσει όλα αυτά τα εργαλεία έχουμε διάφορα μέσα για άμυνα ε, για προστασία πολυμερή εργαλεία ε, εργαλεία θεσμικού χαρακτήρα. Και τέλος, να σας πω, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι προστιθέμενη αξία μπορεί να έχουμε όσον αφορά το έργο που έχει επιτελέσει η Υπηρεσία και η Μογκερίνη για την παγκόσμια στρατηγική μας και για την λευκή βίβλο για την άμυνα. Η προστιθέμενη αξία πρώτα-πρώτα είναι η ρήτρα αναθεώρησης. Προτείνω η αναθεώρηση να γίνεται κάθε πενταετία. Να υπάρχει συντονισμός με το κάθε φορά καινούργιο κοινοβούλιο και την καινούργια επιτροπή. Και έτσι να διαπιστώνεται εάν οι στόχοι και προτεραιότητες ακόμη ε, είναι σύντονες με το περιβάλλον όπου κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, επίσης, θα μπορεί, είπατε εκπρόσωπο και αντιπρόεδρος επιτροπής, να συμμετέχει στην αναθεώρηση. Επίσης, άλλο στοιχείο προσθέμενες αξίες από το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο είναι το Κοινοβούλιο της Ένωσης, οπότε θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, εποπτεία από πλευράς του Κοινοβουλίου επί της εξωτερικής πολιτικής για αυτό το. Ε, επίσης θα πρέπει να ε, στρατεύονται περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια σε κάποιες διαδικασίες διαβούλευσης και έτσι να ενστερνίζονται τις στρατηγικές σε επίπεδο εθνικό. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ένωση των πολιτών επίσης, άρα θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία. Περιμένω πώς και πώς να τα συζητήσουμε σήμερα, να ακούσω τις προτάσεις σας και είμαι ανοιχτή ή στο να λάβω υπόψη όσα θα πείτε και να προσπαθήσω όλα αυτά να τα ενσωματώσω στο σχέδιο κειμένου και σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε Σάντρα, λέει ο πρόεδρος. Και τώρα να αρχίσει η συζήτηση. Για να ακόμη στην Πορτογαλία, είναι η πρώτη και γύρω που έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη συνάδελφό μας Σάντρα Κανιέτε. Πολύ καλή αυτή η βάση για εργασίες και ο τρόπος που συστηματικά τακτοποίησε τους διάφορους τομείς και με τα χαράς να συμβάλλω κι εγώ με κάποια διατύπωση, κάποιο κείμενο συγκεκριμένο για να αναπτύξουμε περαιτέρω κάποια από τα αναφέρθεντα σημεία της εκθέσεως. Νομίζω ότι πράγματι είναι σημαντικότατο να μιλάμε για πολιτική βούληση στη σε αυτή και θα πρέπει να δούμε ότι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η έλλειψη ηγεσία, λόγω της έλλειψης ηγεσίας συνολικά. Δεν αναφέρω συγκεκριμένο όνομα. Βασικός λόγος αυτός για ένας από τους λόγους των προβλημάτων. Εξίσου σημαντικό και το άλλο. Υπάρχουν όρια όσον αφορά την έκταση του κειμένου. Με την υποβολή τροπολογιών θα έχουμε μεγαλύτερη ευκαμψία. Να καλύψουμε και άλλα σημεία. Ενδιαφέρον αυτό θα είναι ίσως χρήσιμη συνεισφορά που θα συμπληρώνει τα όσα θα παρουσιάσει η Φεντερίκα Μογκερίνη. Και τα κράτη-μέλη θα υθετήσουν κάποιες θέσεις στο Συμβούλιο. Σχετικά με αυτό, πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι για διάφορα στοιχεία. Κυρίως όσον αφορά τα μέσα και τα εργαλεία στα πλαίσια της ΣΚΕΠΑ και της ΚΕΠΑ μέσα που διαθέτουμε και που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επαρκώς ή σωστά. Κάποια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα. Φερρυπίν έχουμε αναπτύξει γνώση στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ και οι γνώσεις αυτές θα ήταν χρησιμότατες. Κυρίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ΚΕΠΑ. Όσον αφορά την αναφορά, τις αναφορές τις διάφορες, Μ' αρέσει η αναφορά των νέων απειλών, των νέων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Στον τομέα των συμφερόντων. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να τα υπογραμμίζουμε τα συμφέροντα, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Όσον αφορά τους στόχους, θα μπορούσαμε να έχουμε πιο συγκεκριμένη διατύπωση όσον αφορά τα μέσα προς χρήση για την επιτύχηση των στόχων. Συνεργασία Ευρωπαϊκής Ενώσεως ΝΑΤΟ. Πρέπει να βρούμε καλύτερη ισορροπία. Είναι μια ευκαιρία για μας να επενδύσουμε στην ΚΕΠΑ. Επαφές με τον ΝΑΤΟ και διάρθρωση με τον ΝΑΤΟ όπου μπορούμε αλλά κάποιοι τομεί δεν μπορούν να καλυφθούν τον ΝΑΤΟ, δεν ενδιαφέρεται τον ΝΑΤΟ και πρέπει να αυξήσουμε την άμυνα και ασφάλειά μα. Και χρειάζεται σχετική διατύπωση. Πρέπει να δούμε επίση και εσωτερικέ πτυχέ. Πού βρισκόμαστε. Τι γίνεται με τους ξένους μαχητές. Γιατί απομακρύνονται, απομονώνονται οι νέοι της Ευρώπης που είναι άνεργοι και τους στατολογούν οι τρομοκράτες. Αυτό σχετίζεται με ανόητες πολιτικές που υθετήσαμε και εφαρμόσαμε. Ανεργία, ανισότητες, διακρίσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το λησμονήσουμε αν αντιμετωπίζουμε μια γενική και παγκοσμίου εμβελίας στρατηγική για τη γειτονία, δεν μπορούμε να μιλάμε για μεταναστευτική κρίση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα, αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έχουμε κάτι παραπάνω από υποχρεώσεις, από ηθικές ε, υποχρεώσεις. Έχουμε νομικές υποχρεώσεις. Αυτό δεν θα πρέπει να θάβεται κάτω από το μεταναστευτικό πρόβλημα. Είμαστε σε πολυσχηδή κόσμο. Πρέπει να κινούμαστε βάσει κανόνων για παγκόσμια τάξη, παγκόσμια δικυβέρνηση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα του ρόλου του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι στη σχετική διατύπωση. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Είναι που ελπίζουμε, που δεν θα συμβεί αυτό, της δυνατότητας να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το Συμβούλιο Ασφαλείας ήταν κάτι που πραγματικά υπονομεύει και εμποδίζει την Ευρώπη από το να κάνει τη διαφορά στην παγκόσμια δικυβέρνηση και να κάνει τη διαφορά όσον αφορά το Συμβούλιο Ασφαλείας, να γίνει πιο αποτελεσματικό. Αν προωθήσουμε τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάτι που θα έπρεπε να κάνουμε, μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερο. Ξέρετε ότι έχουμε πολλά προβλήματα, αντιμετωπίζουμε συγκρούσεις στη γειτονιά μας και πέραν αυτής που σχετίζονται τα προβλήματα με την ανεπάρκεια του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τέλος, να πω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τα δικά μας προβλήματα που σχετίζονται με παγκόσμια συστημικά προβλήματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ρόλο μας. Να δούμε πόσο αποκλίνουμε. Η Ένωση πόσο αποκλίνει και πώς προωθεί τη διαφθορά στον κόσμο λόγω ελλείψεως ελέγχου του οικονομικού συστήματος. Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και θα πρέπει να το θέσουμε. Σχετίζεται κατά πολύ με την παγκόσμια κυβέρνηση ή την έλλειψη αυτής. Και πολλά από τα προβλήματα που δημιουργούν την κρίση και σε άλλες χώρες και τις συγκρούσεις άλλες χώρες πρέπει να αντιμετωπιστούν, γιατί αν δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα χτυπήσουν και την πόρτα μας, όσον αφορά τη γειτονιά μας. Να πω σχετικά με αυτό ότι βεβαίως πιστεύω ότι υπέχουμε συγκεκριμένε υποχρεώσει όσον αφορά τη γειτονία. Κατά την άποψή μας, ίσως πρέπει να εστιαστούμε επί του σκοπού, επί των κριτηρίων, όπως τα κριτήρια της Κοπενχάγης, ανεξάρτητα από το αν θα πετύχουμε τη διεύρυνση ή όχι, διότι είναι αμφίδρομος ε, ο δρόμος, εξετάζεται από τους εταίρους. Αλλά η πρόθεση των κριτηρίων σχετίζεται με τις αξίες μας και πρέπει να προωθήσουμε τις, προθυ... τις απαιτήσεις μας για ασφαλέστερο κόσμο, για ασφαλέστερη γειτονιά. Τούτου λεχθέντος με τα χαράς να συνεργαστώ με τη Σάντρα και τους άλλους συναδέλφους και όπως είπα πράγματι έχουμε μια άριστη βάση για ένα κείμενο που θα πρέπει να υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Αλιό Μαρή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Σάντρα για τη δουλειά της που έχουμε συνεργαστεί και από την αρχή μαζί της και άρα δεν έχω πάρα πολλά θέματα να αναφέρω. Η έκθεση αυτή πιστεύω ότι πραγματικά ε, θέτει δύο τύπου ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει και είναι σημαντική με το κατά πόσον η Ευρώπη θέλει να αποτελέσει μια δύναμη όχι μόνο οικονομική αλλά και γεωστρατηγική στο παγκόσμιο προσκήνιο. Και αυτό έχει πάλι δύο υποκατηγορίες. Καταρχάς, η Ευρώπη θέλει να έχει τα μέσα προκειμένου να μπορεί να προασπιστεί την επικράτειά της, η οποία ορίζεται ενδεχομένω επιπλέον με το θέμα της προσχώρησης νέων κρατών, αλλά και να προασπίσει την επικρατειά της, τους πολίτες της και τα συμφέροντά της. Τα συμφέροντά της, τα οικονομικά της συμφέροντα, αλλά όχι μόνο τα οικονομικά συμφέροντα, τα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά συμφέροντα και τα συμφέροντα της ασφάλειας. Πέρα από αυτό, και αυτή είναι η δεύτερη υποκατηγορία, η Ευρώπη έχει να κάνει με, όσα ξεπερνούν την επικρατεία της. Έχει ευθύνη για το παγκόσμιο προσκήνιο για την ανάπτυξη των χωρών, για την δικαιοσύνη, για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς. Και αυτό έχει να κάνει με την ε, ειρήνη στον κόσμο, κατά πόσον θέλει να έχει στη χέρια της τα μέσα. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, αλλά και ένα θέμα μέσων, αν θέλουμε πραγματικά να μπορούμε να δράσουμε. Από αυτή την άποψη λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μία μικρή διασαφήνιση σε ό,τι αφορά τη χρονική, σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ. Είμαστε πυλώνας του ΝΑΤΟ, ο πρώτος εισφορέας σε ό,τι αφορά στρατιωτικές δυνάμεις στο ΝΑΤΟ. Είμαστε ο πρώτος εισφορέας και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Είμαστε λοιπόν το ΝΑΤΟ, αλλά εκ παραλίλου είμαστε και ένας πυλώνας και το θέμα είναι κατά πόσον μπορούμε να προβλέψουμε ειδικέ σχετικές ε, ενέργειες. Αυτό ειλικρινά το πιστεύω. Το ποιε θα είναι αυτές οι ενέργειες θα είναι σίγουρα συμπληρωματικές προς αυτές του ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει να, είπε, να θυμηθούμε και ποιος είναι ο ρόλος μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ένα άλλο δεύτερο θέμα είναι να γνωρίζουμε κατά πόσον θέλουμε να δώσουμε στην Ευρώπη τα απαραίτητα μέτρα μέσα προκειμένου να έχουμε νέες μορφές προάσπισης των, της επικυριαρχίας μας και της λειτουργίας των κρατών μας, κατά πόσον θα δώσουμε τα δομικά και χρηματοδοτικά μέσα. Αν θέλουμε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή άμυνα που να λειτουργεί, θα πρέπει να έχουμε και τα μέσα πρόληψης και πρόβλεψης των κρίσεων και αντίδρασης της κρίσης. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι τίθενται τα πιο μεγάλα ερωτήματα σε ό,τι αφορά την έκθεση της ε, Σάντρα και αυτά θα πρέπει να τα θέσουμε και στους εταίρους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Λούζιν έχει τώρα το λόγο. Θα μιλήσω γερμανικά, σας παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ κυρία Καλνιέτε για το σχέδιο έκθεσης. Να σας ευχαριστήσω εξ αρχής. για το γεγονός ότι το θέμα το οποίο δυστυχώς πάντα παραμελείται, αλλά είναι πολύ σημαντικό, του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια δώσατε μία ξεχωριστή παράγραφο. Εμείς από την ΚΟΕ NGL ε, υποστηρίζουμε το θέμα αυτό και ιδιαίτερως ότι αφορά την εξωτερική πολιτική. Αλλά ο έλεγχος δεν ε, μπορεί να περιορίζεται σε μια υποχρέωση ε, ελέγχου εξωτερικού θα πρέπει να χτιστεί αυτή η σχέση. Στην παράγραφο 15 υποστηρίζουμε επίσης αυτά που αναφέρεται για μια παγκόσμια τάξη και για την παγκόσμια διπλωματία. Αλλά αυτή η διπλωματία θα πρέπει να περιέχει πολλά στοιχεία και οι κανόνες είναι η χάρτα του ΟΗΕ και γενική συνέλευση. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι δεσμευτικοί για όλους λοιπόν τους φορείς. Τι πλέον για την έκθεσή σα. Υπάρχουν διαστάσεις απόψεων και υπάρχουν και διαφορετικές προτεραιότητες από δική μας πλευράς. Είμαστε κατά της ε, μεγαλύτερης ε, στρατιωτικής διάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της απόκτησης εξοπλισμού. Και αυτό έχει να κάνει και με το ΝΑΤΟ. Θεωρούμε ότι είναι παιχνίδι με τη φωτιά αυτό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανατολική διάσταση των δράσεων του ΝΑΤΟ. Το 2% στόχο για τα έξοδα και τα μέσα εξοπλισμών. Είμαστε αντίθετοι. Θεωρούμε ότι είναι λάθος αυτή η κατεύθυνση. Ιδιαίτερα σε καιρού που τα κονδύλια για κοινωνικούς σκοπούς λείπουν. Σε όξυνση των κοινωνικών διαφορών. Στην παράγραφο 8 μιλάτε για τη συνεργασία με τις χώρες της γειτονίας της Ένωσης, ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και να επεκταθεί. Συμφωνούμε. Για να υπάρξει σταθερότητα και ειρήνη. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ένας νέος προσανατολισμός της πολιτικής γειτονίας. Πραγματική υποστήριξη των κοινωνικών και οικονομικών εξελίσεων τέλος στις νεοφιλελεύθερες τάσεις που εξυπηρετούν μόνο τα οικονομικά συμφέροντα της κάθε ελίτ των χωρών και των ομίλων των μεγάλων. Η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία δεν μπορεί να είναι το γεωπολιτικό παιχνίδι της Ευρώπης. Η Άννα Γκόμες μίλησε και για το πόσο σημαντικό είναι να καταπολεμούμε τις αιτίε των διενέξεων. Ε, η ανάλυση αιτίου και αιτιατού στην ευρωπαϊκή πολιτική είναι πάντα μονομερής, πιστεύω. Δεν υπάρχει ανάλυση για το πόσο η ευρωπαϊκή πολιτική προκαλεί ενδεχομένως πιο πολλά προβλήματα από τη λύνη. Η πολιτική των εξωτερικών υποθέσεων θεωρώ ότι προκαλεί ως τώρα πιο πολλά προβλήματα. πολιτική ελεύθερη εμπορία κτλ. για παράδειγμα. Σε αυτά θα περιοριστώ. Συνολικά, ως Αντζιέλ και εγώ προσωπικά Ευρωπαϊκή, ότι η θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει ως διαμεσολαβητής και όχι παρεμβατικά ε, να συνεχίσει να παίζει στρατιωτικό ρόλο. Τέλος, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την έκθεση αυτή θα καταθέσουμε τροπολογίες και ενδεχομένω θα καταθέσουμε και μειονοτική έκθεση. Ευχαριστούμε συνάδελφε Λέζιμ. Και τώρα ο συνάδελφος Μιλανμόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Yo también quiero felicitar a Sandra Καλνίτη por su informe. παρά να συγχαρώ τη Σάντρα Καλνίτη για την έκθεσή τη. στο θέμα το οποίο εδώ έχει αναπτύξει είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να πούμε ότι έρχεται στη σωστή στιγμή γιατί θα δούμε κατά πόσον τώρα ε, ακούγεται η φωνή του Κοινοβουλίου με, με αυτή την έκθεση που έχει τώρα για το Συμβούλιο του Ιουνίου, κυρία Μογκερίνη. Ε, και αυτό επίσης το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι ο στόχος της έκθεσης. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ φιλόδοξο, πολύ πιο φιλόδοξο από αυτά τα ορόσημα τα οποία συνήθως επιβάλλονται σε όλους τους συντάκτες έκθεσης. οπότε λόγω των φραγμών αυτών έπρεπε να δώσει στην κυρία Καλνιέτε, όπως γίνεται και πάντοτε για ε, κάποιου είδους εκθέσεις που έχουν τέτοιες διαστάσεις και προεκτάσεις εγκυκλοπαιδικών, τεραστίων διαστάσεων. Ε, έτσι είναι, έτσι καταλαβαίνω εγώ τα θέματα της άμυνας. Και επίσης όσον αφορά την εξωτερική δράση της Ένωσης, τα θέματα δεν είναι μόνο η άμυνα. Πάμε πολύ παραπέρα. Στην άμυνα βέβαια υπάρχει ακριβώς το έλλειμμα και όπως αντιλαμβάνομαι το Ισλαμικό κράτος αποτελεί μια απειλή. Ή στην Συρία έχουμε τη στάση Ουκρανίας αλλά και Ρωσίας σε σχέση με αυτά. Και ε, τι έγινε επίσης στη Μάλη. Γιατί έχουμε τα θέματα της προστασίας του πολίτη ε, τα οποία έτυχαν προτεραιότητος ή στην έκθεση. Και άρα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια στρατιωτική συμμαχία. Ούτε και αρα θα πρεπει να συνειδητοποιησουν την ευρωπαικη ενωση δεν ειναι μια στρατιωτικη συμμαχια ουτε και σκοπευουμε να την κάνουμε τέτοια. Είδατε, είναι πολύ πιο Για κοιτάξτε το άρθρο 3, παράγραφος 5 τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί που λέει για τους στόχους Ευρωπαϊκή Ένωση στα εξωτερικό. Ε, όχι, δεν επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά ή στην προστασία των πολιτών, όπω το είπε και η Σάντρα Καλνιέτε. Έχουμε τα συμφέροντα, έχουμε τι αξίε, τι αρχέ, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εξωτερικό εμπόριο, όλα αυτά και αυτό θα πρέπει να αποφύγουμε είναι να μην δοθεί λάθος εντύπωση από την έκθεση. Ότι δηλαδή θέλουμε με την έκθεση να δώσουμε βάρος άνισο, υπέρ της άμυνας. Προσοχή της προτεραιότητας, γιατί πρώτα για να είμαστε πρώτα-πρώτα ε, παίκτης, πρέπει να είμαστε πρώτα-πρώτα πρωταγωνιστής και παίκτης παγκόσμιος και όχι περιφερειακός. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει από την ενημερία όμως και στην γειτονιά μας. Εγώ είμαι μεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι ε, εκφύσεως της είναι παίκτη παγκόσμιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε υπάρχουν ε, κράτη-μέλη τα οποία ανήκουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και άλλοι που δεν είναι μόνιμα μέλη αλλά έχουν όπως η χώρα μου η Ισπανία ε, ακτινοβολία παγκόσμια δηλαδή ότι επηρεάζουμε τα τεκτενόμενα στην Λατινική Αμερική. Α, και η Πορτογαλία επηρεάζει και κράτη της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Άρα δεν μπορούμε να ε, περιοριστούμε ως Ευρώπη μόνο εδώ στη γειτονιά μας. Έχουμε βέβαια και το εξωτερικό εμπόριο το οποίο αφορά όλες τις χώρες του κόσμου και έχουμε βέβαια από την άλλη μεριά την εξάρτησή μας τον υπόλοιπο κόσμο με τις πρώτες ύλες. που μας αφορούν όλα όσα γίνονται παντού στον κόσμο. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε στην πολιτική μας φιλόδοξη και παγκοσμίων διαστάσεων. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βάλουμε όλα εδώ, ούτε καν τα οικονομικά και γι' αυτό αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Κανιέτε ε, είναι αγκάστη να δώσει κάποιε συγκεκριμένε προτεραιότητε. Όμω νομίζω ότι σε τέτοιου είδου εγκυκλοπαιδικών διαστάσεων εκθέσει είναι δύσκολα τα πράγματα και δεν είναι δυνατόν να, να, να, να τα βάλουμε μέσα στο στενό κορσέ των, των συγκεκριμένων λέξεων. Αυτά δηλαδή που μας επιβάλλει η γραμματεία. Εγώ θα βάλω την τροπολογιούλα μου σαν λιθαράκι και έτσι νομίζω ότι θα διευρύνω κάπως το βελνικέ της έκθεσης. Αλλά, αλλά σας ξαναλέω το έργο της ε, συντάκτριας ήταν τόσο περιορισμένο από αυτό τον κορσέτο των συγκεκριμένων γραμμάτων και λέξεων και σελίδων. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι κάνει ε, όχι μόνο η εξωτερική πολιτική ένωση, τι κάνει στο εμπόριο, στο περιβάλλον, στην οικονομία. Δύσκολα, δύσκολα αυτά. Μπράβο στην κυρία Καρδινιέτε. Την ευχαριστώ, τη συγχαίρω. Οπότε και επιτρέψτε μου να αποπειραθώ και εγώ με την τροπολογιούλα μου να βάλω ένα και Ευχαριστώ. Thank you ε, Εμείς σας ναι. ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι είναι κρίμα που τόσο σημαντική έκθεση για την οποία δώσαμε τόσες μάχες στο Προεδρείο και ήταν και η δια πρωτοβουλία της Επιτροπής μας. Γιατί να μην έχουμε τώρα να τη συζητούν τόσο πολλούς βουλευτές. Αυτό είναι το πλαίσιο του έργου μας στους επόμενους μήνες και από πλευράς μου θεωρώ ότι είναι σημαντικό να δούμε το πώς θα έχουμε ε, την ολοκλήρωση της οικοδόμησης και το state building στην Ευρώπη και έτσι είπαμε ότι πάμε για τις εκλογές με τα συγκεκριμένα εργαλεία ούτως ώστε να μπορέσουμε να κοντράρουμε τις, όλες τις, τα θεσμικά όργανα, τα παγκόσμια ε, και έτσι ε, να μπορέσουμε να ενεργήσουμε και προς την κοινωνική πλευρά για την φτώχεια και να έχουμε τις μεταρρυθμίσεις, να φροντίσουμε τα σύνορα, τις μαφίες, τους μετανάστες. Να δούμε τι θα γίνει με τη διαχείριση των, των συγκρούσεων συγγνώμη, και να δούμε και το περιβάλλον, τι γίνεται με τις, με τις νάρκες, τι γίνεται με τους αφοπλισμούς. Αγαπητή Σάντρα, σε ευχαριστούμε για την έκθεση, αλλά ευχαριστούμε και όλους όσους συνέβαλαν. Οπότε τώρα να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση με παρεμβάσεις και να σας πω και πότε είναι και η προθεσμία για τις τροπολογίες. Καλνιέται. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους ε, όσους ε, εξέφρασαν σε για το σχέδιο εκθέσεως. Ε, δεν θα σταθώ σε αδίποτε προτασίες σας αναμένω να καταφθάσουν υπομορφήν τροπολογιών της εκθέσεως. Και όπως προανέφερα, είμαι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις. Πραγματικά θέλω να συμπεριλάβω ό,τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Θέλω μια ισορροπημένη έκθεση, το κείμενο να είναι στεναρό. Ξέρετε το σχέδιο κειμένου έχει κάποιο συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων γραμμάτων που περιλαμβάνει και γι' αυτό εγώ πρόβαλα τα σημαντικότερα ζητήματα. Όλοι μαζί μπορούμε να καλύψουμε αυτά που αισθάνεστε που πρέπει να καλύψει η έκθεση και τα οποία δεν εκάλυψε. Τα διάφορα κενά τα καλύψουμε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάντρα. Λοιπόν, για σας που παρίσταστε προθεσμία για τις τροπολογίε είναι 22 Φεβρουαρίου, που σημαίνει ακριβώ σε λιγότερο από μια εβδομάδα από σήμερα θα ψηφίσουμε την έκθεση στις 15 Μαρτιού εδώ στην Επιτροπή και αναμένεται στην Ολομέλεια 11 με 14 Απρίλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταφέραμε να τηρήσουμε το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για σήμερα. Σας ευχαριστώ. Την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό σας βράδυ.